Good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι ιδιαίτερως που σας ξαναβλέπω σήμερα το πρωί και ελπίζω χθε να καταφέρατε να ήρθατε στις Βρυξέλλες. Το δικό μου ταξίδι προς Βρυξέλλες ήταν πολύ ενδιαφέρον. Χρειάστηκε να ταξιδέψω 14 ώρες για να φτάσω μέχρι τις Βρυξέλλες λόγω του μεγάλου χάους που επικράτησε στις ε, αεροπορικές εταιρείες και σε αεροπορικές μεταφορές. Πάντως ευχαριστώ για την, για την κατανόησή σας. Σήμερα ξεκινάμε την κατάμεστη ημερήσια διάταξή μας με τις ψηφοφορίες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την ψηφοφορία της έκθεσής μας ε, με θέμα την πολιτική συνοχή και την κυκλική οικονομία. Ο εισηγητής μας είναι ο κύριος Σκύρλετς. Δεν ξέρω αν θέλετε το λόγο κύριε εισηγητά πολύ σύντομα να ευχαριστήσω τους και όλους για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Ωραία. Οπότε πάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Ξεκινάμε με την τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ? κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 7 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 13 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 15 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 17 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 17 Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 30 λέει η πρόεδρος λάθος, λάθος ε, συγγνώμη λέει η πρόεδρος η 30 καταπίπτει και πάμε στην 32 ποιος είναι υπέρ υπέρ της 32 δεύτερο τμήμα ή μάλλον πρώτο τμήμα από την αρχή. Τροπολογία 32, πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 32. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 33. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 38. Ποιος είναι υπέρ Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Ποιος είναι υπέρ. Αν από τη στιγμή που εγκρίναμε την τροπολογία 42, η τροπολογία 12 της Επιτροπής Περιβάλλοντος καταπίπτει. Γι' αυτό πάμε στην 5. Περ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία 5. Τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 51. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 58. Ποιος είναι υπέρ? Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 59. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 60. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 61. Έχουμε μια προφορική τροπολογία. Είναι κανείς κατά τις προφορικές τροπολογίες. Όχι. Οπότε ψηφίζουμε την τροπολογία 61 μαζί με την προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 67. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 71. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην συμβαστική τρο... μάλλον στην τροπολογία 79. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 11. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 82. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 90. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 91. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 92. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 103. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 104. Υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 105. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 110. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 111. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 112. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 113 μαζί με την προφορική τροπολογία. Είναι κανείς κατά της προφορικής. Όχι. Οπότε ψηφίζουμε την 113 μαζί με την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 124. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 19. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 127. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 20. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 131. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 6 της έμβη υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Έμβη 7 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Έμβη 8 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Έμβη 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. MV10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. MV13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. MV16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. MV17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. MV18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. MV19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. MV20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. MV22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας και η έκθεση εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Σκέρλετς. Οφείλω να πω ότι έχουμε μία επιπλέον θετική ψήφο του εισηγητού που ξέχασε σήμερα την ηλεκτρονική κάρτα ψηφοφορίας. Την προσθέτουμε. Ε, συμβαίνουν κύριε Σκέρλετς αυτά. Και περνάμε στο επόμενο θέμα. Ψηφοφορία για τη γνωμοδότησή μας «Ρόλος των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης». Γνωρίζετε ότι την έκθεση την επονεί η Επιτροπή ΑΦΚΟ και ο κύριος Όλμπριχτ έχει συντάξει τη δική μας γνωμοδότηση για την έκθεση. Κύριε Όλμπριχτ, θέλετε το λόγο? Δεν είναι εδώ σήμερα. Ε, πάμε απευθείας στην ψηφοφορία. Ξεκινάμε με τη συμβαστική υπαριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 30, ε, συγγνώμη, τροπολογία 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε την γνωμοδότηση όπως τροποποιήθηκε, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, εγκρίνεται με 30 ψήφους υπέρ. 30 συν 1. Ε, τελειώνει και αυτή η γνωμοδότηση και πάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία. Ψήφισμα εκ μέρους της Επιτροπής της δικής μας για τις συγκεκριμένες ανάγκες των ε, ορεινών και απόμακρων περιοχών της υπαίθρου. Πρωτού ψηφίσουμε, πρέπει να σας αναγγείλω ότι αποφασίσαμε να συντάξουμε αυτό το ψήφισμα στις 25 Απριλίου. Ε, τότε συμφώνησαν οι συντονιστές να στηρίξουν το σχέδιο ψηφίσματος και το σχέδιο μοιράστηκε στα αγγλικά στα μέλη της Επιτροπής Ρέντζη μέσω της γραπτής διαδικασίας και λάβαμε 42 τροπολογίες πριν λήξει η προθεσμία. Τώρα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ποια θα είναι τα επόμενα στάδια της διαδικασίας. Οι συντονιστές θα συντάξουν ερώτηση βάσει του άρθρου 128 ε, του εσωτερικού κανονισμού. Θα συντάξουν λοιπόν προφορική ερώτηση που θα υποβληθεί εκ μέρους της Επιτροπής μας για να λάβουμε απάντηση. Αν οι πολιτικέ ομάδε συμφωνήσουν να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη η ερώτηση αυτή, θα συζητηθεί το θέμα στην Ολομέλεια. Με αφορμή την ερώτηση και μετά και του ψηφίσματο. Αυτό ήθελα να σα υπενθυμίσω. Και τώρα δεν έχω εγώ να πω κάτι. Ευχαριστώ όλους για τις συνεισφορές τους την σύνταξη του ψηφίσματος και για την ε, πολύ δραστήρια συμμετοχή τους στι τροπολογίε και στην εξέβριση συμβαστικών λύσεων. Ε, τροπολογία 3 με προφορική τροποποίηση. Είναι κανείς κατά της προφορικής τροπολογίας. Ωραία, ψηφίζουμε την τροπολογία 3 λοιπόν. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 με προφορική τροπολογία πάλι. Είναι κανεί κατά τη προφορική τροπολογία, όχι. Τροπολογία 4 λοιπόν με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Επιτρέψτε μου να κάνω εδώ μια προφορική τροπολογία διότι η δεύτερη πρόταση στη συμβαστική άλλαξε χθε το βράδυ και θα λέγεται εφόσον πολλοί πολίτε σε αστικά κέντρα θα πρέπει να έχουν την εξασφάλιση ότι απολαμβάνουν ε, παρόμοιες ευκαιρίες με αυτούς που ζουν ε, στις περιοχές της Πέθρου. Αυτό είναι το συμβαστικό κείμενο. Ναι, ναι εάν μου επιτρέπετε αυτό καλύπτει τώρα και τις τροπολογίες 10 και 11 η συμβαστική. Οπότε όχι απλώς καλύπτει την αιτιολογική σκέψη Ή e, αλλά και G. Ε και Εάν εγκριθεί αυτή η συμβαστική. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, σκόπευα να το πω και από μόνη μου. Διότι το συζητήσαμε με την γραμματεία. Διότι αυτή η συμβαστική καλύπτει μια σειρά από άλλες τοπολογίες Τροπολογία 7, 10, 11 και 31. Πρόκειται για τροπολογίες που όλες έχουν σχέση με την ατολική σκέψη G. Άρα η συμβαστική ανακαλύπτει τον αιτιολογική σκέψη ε και σ, όπως είπε ο συνάδελφος. Με όλες αυτές λοιπόν τις προφορικές τροπολογίες και όλες αυτές τις διευκρινήσεις για τις αιτιολογικές σκέψεις, ποιος είναι υπέρ της συμβαστικής υπαριθμών 1. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίφθηκε, αλλά καλύτερα να το ελέγξουμε. Τροπολογία 8. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ ψηφίστε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτής. Εγκρίνεται. Κύριε Σκρέτς. Ναι. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Η 9 καταπίπτει. Πάμε στην 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, καταπίπτει. Με συγχωρείτε, κατέπεσε. Η 14 κατέπεσε. 15 με προφορική τροποποίηση. Είναι κανεί κατά τη προφορική, όχι. Ωραία, λοιπόν, υπέρ με την προφορική τροπολογία. Κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Α, καταπίπτει, καταπίπτει. Η 37 εγκρίθηκε, οπότε καταπίπτει η 38. 39, ε, 41, συγγνώμη, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 42, 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική, άρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται το ψήφισμα. 31 ψήφι υπέρ. 31. Ευχαριστώ πολύ. Here we close our voting time. Και ολοκληρώσαμε τις προφορίες μας στην ώρα μας. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε ακάθεκτη. Και τώρα να συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Εξέταση του σχεδίου έκθεσης. May I ask the members who are... Παρακαλώ όσοι συνάδελφοι φεύγουν από την αίθουσα να το κάνουν αυτό σιωπηρός. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε λοιπόν με το επόμενο σημείο στην εμμυρίσια διάταξη. Είναι η εξέταση της έκθεσης, του σχεδίου έκθεσης. του ε, εισηγητή μας, του κυρίου Αριμού, ειδικά μέτρα για την Ελλάδα βάσει του κανονισμού 2015-1839. Σας παρακαλώ οι σύμβουλοι από τις ομάδες να σταματήσουν ε, τα πηγαδάκια. Χρειαζόμαστε ησυχία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ρημό, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα θα μια σύντομη παρουσίαση της έκθεσής μου, έτσι όπως το έκανα και πριν από δύο εβδομάδες. Θα σας Πρόκειται για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ε, Επιτροπής Περιφερειακής ε, Πολιτικής για τα σχέση ειδικά μέτρα για την ε, Ελλάδα βάσει του κανονισμού 2015 κάθετο κάθετος 1839 και θα ήθελα ως προημίου να πω ότι δεν πρόκειται για μία συζήτηση εν σχέση με τα αίτια αυτών των έκτακτων μέτρων γιατί η Ελλάδα απέλθε σε αυτή την κατάσταση, αλλά η έκθεσή μου πραγματεύεται το θέμα, το ζήτημα των επιπτώσεων αυτών των ειδικών μέτρων, κατά πόσον αξιολογούνται θετικά αρνητικά, κατά πόσο έχουν, μπόρεσαν να ολοκληρωθούν τα προγράμματα μέσω αυτών των δύο μέτρων ή όχι. Και αντιστοίχω, ε, θα προβώ μια πολιτική αξιολόγηση των... Δεν θα προβώ μια πολιτική αξιολόγηση των λόγων για το ξέσπασμα της κρίσης ε, και επίσης και εσείς δεν θα έπρεπε να ε, τοποθετηθείτε σε σχέση με τα αίτια της κρίσης. Λοιπόν, περί τίνος πρόκειται. Η Επιτροπή το 2015 ορθά αναγνώρισε ότι η Ελλάδα λόγω της ε, κατάστασης στην οποία είχε βρεθεί λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης δεν μπορούσε να διαθέσει τα χρήματα για προγράμματα στο πλαίσιο Ταμείου Συνοχής ή Περιφερειακής ε, Ανάπτυξης προκειμένου να ελοπίσει κάποια σχετικά προγράμματα, δηλαδή να καλύψει το δικό της ποσοστό της συγχρηματοδότησης αυτών των προγραμμάτων. Και η Επιτροπή πρότεινε να ληφθούν δύο ειδικά μέτρα προκειμένου να βοηθηθεί η Ελλάδα. Πρώτον, ε, για, την, ε, για τα προγράμματα που μπήκαν στην περίοδο 2007-2013 το ποστό συγχρηματοδότηση τη Ελλάδα καταργήθηκε. Έτσι λοιπόν χορηγήθηκε μια χρηματοδότηση 100% εκ μέρου τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο οδήγησε με πλέον ρευστότητα τη τάξη του ενό δις δισεκατομμυρίου ευρώ ή θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτό. Και το δεύτερο ειδικό μέτρο ήταν ότι για την περίοδο 2014-2020 μια πρώτη προχρηματοδότηση ε, χορηγήθηκε, θα έπρεπε να χορηγηθεί νωρίτερα, ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Έτσι λοιπόν ο συνολικός όγκος ήταν περίπου δύο δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα. Και όπω αναφέρθηκε στον τίτλο, πρόκειται για ένα ειδικό μέτρο στο πλαίσιο τη απλουστευμένη διαδικασία. Αποφασίστηκε εδώ στο Κοινοβούλιο για ένα απλό λόγο, γιατί ήταν κατεπίγουσα η χορήγηση αυτή τη βοήθεια, γιατί η Ελλάδα έπρεπε να ολοκληρώσει αυτά, να ελοπίσει αυτά τα προγράμματα και γι' αυτό αυτά τα δύο δι, υπό την έννοια αυτή τα χρειαζόταν κατεπηγόντως. Στον κανονισμό αναφέρεται ότι η Ελλάδα μέχρι το Δεκέμβριο του 2016 ε, έπρεπε να καταθέσει μια έκθεση. Το γεγονός ότι τώρα το 2018 βρίσκομαι εδώ και όχι το 2017 για να κάνω την έκθεση για τα ειδικά αυτά μέτρα οφείλεται στο ότι η Ελλάδα δεν εκπώνησε την έκθεση αυτή τα τέλη του 2016 αλλά το Μάιο του 2017 και η Επιτροπή δεν ε, διαβίβασε την ε, έκθεση αυτή στο Κοινοβούλιο παρά τις επανειλημμένες ε, αιτήσει και προφορικές προφορικά ερωτήματα τα οποία υποβάλαμε και ενώ εγώ χρειαζόμουν την έκθεση αυτή προκειμένου να κάνω αυτή την αξιολόγηση γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτή η καθυστέρηση του ενός έτους. Στο σχέδιο έκθεσής μου ε, έκανα και μία αξιολόγηση και μπορούμε να καταλήξουμε στο εξή. Αυτή η επιπρόσθετη ρευστότητα πράγματι αξιοποιήθηκε αποτελεσματικά εκ μέρου τη Ελλάδα προκειμένου πράγματι να ολοκληρωθούν πολλά προγράμματα και αυτό μπορούμε να το αναφέρουμε και με αριθμού. Η Ελλάδα στην περίοδο αυτή ε, ε, δούλεψε πάνω σε έναν κατάλογο προγραμμάτων ε, προτεραιότητων, κατάλογος 161 προγραμμάτων τα οποία αφορούν 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2007-2013. 55% ε, όλων των προγραμμάτων από αυτά τα 136 ολοκληρώθηκαμε το τέλο του 2017. 27 από αυτά τα προγράμματα προτεραιότητας μεταφέρθηκαν στην επόμενη περίοδο 2017 με 2020 και ένα πρόγραμμα ε, και ορισμένα προγράμματα που αφορούν 1,1 δις δεν συνεχίστηκαν και διακόπηκαν. Όσο πρόγραμμα για τα πετυχημένα προγράμματα, τα λεγόμενα προγράμματα γέφυρα από την προηγούμενη ε, περίοδο 2000-2006 και συνέχισαν ε, και ολοκληρώθηκαν μάλλον στην περίοδο 2007-2013, μπορούμε να αναφέρουμε κάποιους αυτοκινητοδρόμους οι οποίοι ανακαινίστηκαν, το μετρό στην Αθήνα, το μετρό στη Θεσσαλονίκη και την σιδηροδρομική σύνδεση ε, μεταξύ τη Θωρέας, Λιανοκλαδίου και Δομοκού. Προγράμματα τα οποία λόγω αυτών των ειδικών μέτρων πράγματι υλοποιήθηκαν και εγώ το εξακρίβωσα και εάν δεν είχαν ληφθεί αυτά τα ειδικά μέτρα ως Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, τα προγράμματα αυτά δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν και αυτό θα είχε σαν συνέπεια το ελληνικό κράτος να πρέπει να διακόψει ε, αυτά τα προγράμματα γιατί θα έπρεπε να τα είχε χρηματοδοτήσει μόνο του. Και αν δεν είχε τα χρήματα αυτά της, ε, και θα έπρεπε να επιστρέψει τα χρήματα αυτά της προ-χρηματοδότηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα οδηγούσε μια περαιτέρω όξυνση της κρίσης. Στη νέα περίοδο ε, ενίσχυσης ε, έχουμε, έχουν οριστεί 18 προγράμματα προτεραιότητας τα οποία λόγω της προχρηματοδότησης ε, έχουν ξεκινήσει, υπάρχουν δύο αριθμοί που θα πρέπει να αξιολογήσουμε θετικά το πρώτο είναι σημαντικό νούμερο, ότι τα ποσοστά απορρόφησης για την περίοδο 2007-2013 είναι 100%, δηλαδή τα κονδύλια τα οποία δόθηκαν στην Ελλάδα πράγματι εισέρευσαν στα προγράμματα αυτά και αυτή ήταν μια προϋπόθεση για την χορήγηση της χρηματοδότησης και υπάρχει και ένα δεύτερο νούμερο το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί θετικά. Τα ποσοστά απορρόφησης για την περίοδο 2014-2018 είναι 28% ή 23% όπως λέει η Επιτροπή, δηλαδή είναι τα ανώτατα όρια του μέσου στην Επιτροπή. Και ένα τρίτο νούμερο που θα πρέπει να αναφέρουμε Λόγω της ε, προηγούμενης ε, περίοδου και των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στην περίοδο αυτή, το ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2% από ό,τι θα είχε αυξηθεί ε, χωρίς τα χρήματα αυτά, κάτι το οποίο είναι σημαντικό για την ανάπτυξη της Ελλάδας. Τελική παρατήρηση, πως τα απορρόφηση και ΑΕΠ είναι δείκτες οι οποίοι μας λένε κάτι τόσο για την ποσότητα, σε ποσοτικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο των οικονομικών, αποτελε... οικονομικών στοιχείων. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει κατά πόσο τα προγράμματα αυτά επίσης καθορίζονται από το στοιχείο της ε, ποιότητας. Αλλά διαπιστώνουμε ότι τα χρήματα αυτά πράγματι χρησιμοποιήθηκαν ε, δεν ε, τελμάτωσαν τα προγράμματα αυτά, ούτε διακόπηκαν, διακόπησαν. Άρα λοιπόν ε, θα πρέπει να αύξησαν υπό την έννοια αυτή και το βαθμό ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Δημιουργήθηκαν θέσεις απασχόλησης και βελτιώθηκαν οι συνθήκες διαβίωσης των Ελλήνων πολιτών. Οι μετέπειτα αναλύσεις θα δείξουν βεβαίως σε ποιο βαθμό ε, τα ειδικά μέτρα αυτά συνέβαλαν ε, θετικά. Η έρευνα αυτή περιλαμβάνει μόνο έναν ε, κατάλογο των προγραμμάτων τα οποία έχουν υλοποιηθεί, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να πούμε αν κατακλείδη ότι πράγματι ήταν η απολύτως ορθή απόφαση να ληφθούν αυτά τα ειδικά μέτρα στο πλαίσιο του εν κανονισμού. Και δεν βοηθήσαμε μόνο την Ελλάδα, με τα μέτρα αυτά δεν ε, βάλαμε χρήματα σε προγράμματα τα οποία έχουν μια υπεραξία για την Ελλάδα και την Ευρώπη αλλά επίσης εμποδίσαμε πολλά χρήματα ε, να χαθούν με τη μη υλοποίηση των προγραμμάτων και επίσης εμποδίσαμε και την επιστροφή των χρημάτων αυτών στην Ευρώπη, κάτι που θα επιδίνωνε περαιτέρω την κατάσταση της Ελλάδος και θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι πολύ σημαντικό εμείς ως Κοινοβούλιο να αξιολογήσουμε, ε, να προβούμε σε μια αξιολόγηση των ειδικών μέτρων. Δηλαδή δεν θα πρέπει να είναι ε, ένα κανόνα, να καταργεί το συν χρηματοδότηση, αλλά θα πρέπει να αποτελεί μια εξαιρετική περίπτωση παρόλο που στην ελόγω περίπτωση της Ελλάδος, όπως σας είπα, η απόφαση ήταν σωστή. Και θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι είναι σημαντική και στοχευμένη απόφαση να ληφθούν αυτά τα ειδικά μέτρα για την Ελλάδα. Και θα ήθελα με ευχαρίστηση, με μεγάλη ευχαρίστηση να συζητήσω μαζί σας το θέμα αυτό και τις Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Ρήμο. Και τώρα λόγω στους και ηγητέ. Ξεκινούμε με τον κύριο Κοτσολίνο. Πολύ γρήγορα δύο παρατηρήσεις. Θα συμφωνήσω γέννη με την έκθεση και τις προτάσεις της. Απλώς η πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι τα πήγαμε καλά. Τα Ήταν καλή απόφαση να απελευθερώσουμε αυτά τα κονδύλια και να ξεπεράσουμε τις δεσμεύσεις της συγχρηματοδότησης. Ήταν μια επιλογή που είχε θετικές επιπτώσεις και για την ελληνική οικονομία που από τη σκοπιά της υλοποίηση έργων βοήθησε και επίσης έδωσε μια όθηση στην Ελλάδα να είναι το κράτος που χρησιμοποιεί περισσότερο από όλους το, τα κοινοτικά κονδύλια για την περίοδο 2014-2017. Η δεύτερη παρατηρήσή μου είναι ότι ίσως πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από το ιδεολογικό πλαίσιο της συγχρηματοδότησης. Μας ε, περιορίζει πολύ και βλέπω ότι περιορίζει και στην όλη συζήτηση για την νέα περίοδο προγραμματισμού. Διότι τουλάχιστον από την σκοπιά της Ελλάδας μπορούμε να πούμε ότι η πρακτική εμπειρία που είχαμε δείχνει πόσο η συγχρηματοδότηση ε, σχετίζεται με τις πραγματικές δαπάνες και πόσο έχει να κάνει με την πραγματική διάρκεια υλοποίηση των έργων. Επ' αυτού πρέπει να σκεφτούμε. Αυτό είναι μάλλον το πιο ε, ενδιαφέρον όλης της έκθεσης. Και εκεί χρειάζονται περιττέρω διευκρινήσεις από την πλευρά της Επιτροπής και του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Διότι εν απουσία ε, είχαμε επιτάχυνση και ποιότητα στις δαπάνες σημαντικότερη. Τι όρια λοιπόν, τι προβλήματα είναι αυτά που ξεπεράστηκαν και αντιμετωπίστηκαν με την απουσία της συγχρηματοδότησης και έγιναν οι δαπάνες ε, και πιο αποτελεσματικές και πιο γρήγορες. Πρέπει λοιπόν λίγο να ξεφύγουμε από την ιδεολογική δέσμευση της συγχρηματοδότησης και να δούμε τι συνέπειες είχε τελικά αυτή η επιλογή που εντάξει είχε τα ειδικά χαρακτηριστικά, ε, οφειλόταν σε ειδικέ ανάγκες με όλα αυτά που αναφέραμε, αλλά σίγουρα ίσως μας, ε, μας υποδεικνύει μια κατεύθυνση, ένα δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για το μέλλον. Thank Σας ευχαριστούμε εκ μέρους της ομάδα CCR. Ο κύριος Κοζουόφσκι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Φυσικά συμφωνώ με τους ε, δύο προλαλήσαντες σε ό,τι αφορά την ελληνική κρίση. Η κατάσταση στην Ελλάδα απέτησε τη λήψη ειδικών έκτακτων μέτρων και χαίρομαι που ε, αντέδρασε σωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκεκριμένα μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτή την προβληματική κατάσταση. Προβληματική κυρίως για την Ελλάδα αλλά και για τις ε, χώρες της περιφέρειας τις γειτονικές, αλλά και γενικώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν πολύ σημαντικές όλες αυτές οι επιχειρήσεις που έγιναν. Βέβαια, αυτή την αντίδραση θα πρέπει να την θεωρήσουμε ως κάτι απολύτως έκτακτο, εξαιρετικό. Δεν θα πρέπει να είναι συνηθισμένο να κινητοποιούνται τόσο υπέρογκα ποσά σε παρόμοιες καταστάσεις. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν χρειάστηκαν αυτή τη φορά. Όντω ήταν απαραίτητα αυτή τη φορά, αλλά να αναγνωρίσουμε τον ε, εξαιρετικά έκτακτο χαρακτήρα αυτή τη αντίδραση. Ε, σίγουρα η κατάσταση στην Ελλάδα απέδειξε ότι τα κονδύλια που κινητοποιήθηκαν συνέβαλαν στην αναζωγόνηση της ελληνικής οικονομίας και στην αναχέτηση αυτής της ανησυχητικής ε, ε, πορείας της ελληνικής κρίσης. Και εν κατακλείδη θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τη γνώμη του εισηγητού, του κυρίου Αριμού. Ότι δεν γίνεται ε, ποσοτική, ε, ε, ποιοτική μάλλον αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της κατάστασης. Καλό θα ήταν να είχαμε και αυτές τις πληροφορίες και τη ποιοτική αξιολόγηση για τους επιμέρου τομείς για να δούμε όλες, όλα αυτά τα μέτρα, όλε αυτές οι δραστηριότητε ε, ε, κατέληξαν σε κάποια ποιοτική αναβάθμιση. Καλό θα ήταν είχαμε και αυτά τα στοιχεία για να κάνουμε μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση. Ευχαριστώ κύριος Παπαδημούλης, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι η δουλειά που έχει κάνει ο εισηγητής μας, ο κύριος Αριμών, είναι θετική την προσεγγίζω και εγώ προσωπικά και η πολιτική μου ομάδα με θετικό πνεύμα και σκοπεύουμε με την ίδια επικοδομητική διάθεση να καταθέσουμε και ορισμένες τροπολογίες. Η έκθεση που συζητάμε σήμερα δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι κάναμε καλά κυρία Πρόεδρε, κυρία Μιχαήλοβα, που με δική σας εισήγηση φέραμε στην Ολομέλεια για έγκριση τον κανονισμό 1839 το 2015. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία αυτήν την ειδική ρύθμιση και η εξέλιξη και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Ελλάδα τα κατάφερε. Και νιώθω και ως Έλληνας μια ικανοποίηση γιατί στην σωστή απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου που περίπου ομόφωνα ενέκρινε αυτό τον κανονισμό ήρθαν οι ελληνικές αρχές, η ελληνική διοίκηση με τα αποτελέσματα που μας παρουσίασε ο κύριος Αριμών και το Δεκέμβριο μας παρουσίασε και η DG Regio της ε, Κομισιόν να δείξει ότι ολοκληρώθηκαν έργα, βελτιώθηκε η ικανότητα προγραμματισμού και διαχείρισης στην αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων και Θέλω να υπογραμμίσω κάτι, το είπε ο κύριος Σαριμών, η Ελλάδα βρίσκεται πρώτη μέσα στη λίστα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απορρόφηση αυτή την περίοδο. Το είπε και ο κύριος Κοζολίνο. Και αυτή η ευρεία συνένεση όλων των πολιτικών ομάδων στη διαπίστωση των αριθμών και της πραγματικότητας είναι κάτι θετικό όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για τις πολιτικές συνοχής και για τους στόχους που επιδιώκει και η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής. Διότι φαίνεται ότι αυτά τα χρήματα δεν είναι πεταμένα λεφτά. Αντίθετα, αυτές οι ρυθμίσεις βόηθησαν, όπως σωστά είπε ο κύριος Σαριμών, να μην χαθούν λεφτά. Γιατί θα χανόντουσαν χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων αν τα έργα αυτά μέναν μισοτελειωμένα και επομένως άχρηστα, χωρίς καμία θετική επίδραση στην παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την αύξηση των επενδύσεων, τη συμβολή στην άνοδο του ΑΕΠ. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που στην Ελλάδα έχει αρχίσει μια ανάκαμψη. Στις 20 ε, Αυγούστου η Ελλάδα βγαίνει από τα προγράμματα οικονομικής υποστήριξης, τελειώνει με τα μνημόνια και νομίζω ότι η έκθεση που συζητάμε είναι μια ιστορία επιτυχίας και για το Ευρωκοινοβούλιο και για την πατρίδα μου την Ελλάδα και για την Κομισιόν που εισηγήθηκε αυτή την αλλαγή στον κανονισμό. Ως έκτακτη ρύθμιση και όχι ως κανόνα, συμφωνώ και μας δίνει τη δυνατότητα να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα διαχειριστικό και σας το λέω όχι με ιδεολογικά κριτήρια αλλά ως μηχανικός που έχει ασχοληθεί με συγχρηματοδοτούμενα έργα. Γιατί βρεθήκαμε στα χρόνια του 2015 με πάρα πολλά μισοτελειωμένα έργα της περίοδου 2007-2013 με κίνδυνο να καταρρεύσουν αυτά τα έργα και να μην ολοκληρωθούν ποτέ και να χαθούν τα χρήματα διότι δεν έγινε σωστός σχεδιασμός και προγραμματισμός. Και ενώ μπορούσαν να υλοποιηθούν και να τελειώσουν 100 έργα, μπήκαν τα προηγούμενα χρόνια 180 που ήταν αδύνατο να υλοποιηθούν με αυτά τα χρήματα. Άρα μέσα από την ιστορία αυτή βγαίνουν και συμπεράσματα για την ανάγκη ορθολογικής αξιοποίησης των πόρων με ευθύνη και των περιφερειακών αρχών και των εθνικών αρχών και των κοινωνικών αρχών. Καταλήγω ε, με μια πρόταση. Επειδή η έκθεση που συζητάμε καταγράφει ένα θετικό αποτέλεσμα, όπως το περιέγραψε ο κύριος Αριμών, που είναι προϊόν συνεργασίας και συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Κομισιόν και της, των ελληνικών αρχών, προτείνω ο Υπουργός ο Αρμόδιος της ελληνικής κυβέρνησης, ο κύριος Χαρίτσης, να κληθεί, κυρία Πρόεδρε, τον Ιούλιο σε μια προγραμματισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής για να συζητήσουμε όλα αυτά ως ένα παράδειγμα καλής πρακτικής. Και το χρειαζόμαστε γιατί αυτή την περίοδο γίνεται και μια μεγάλη συζήτηση και μια μεγάλη αντιπαράθεση να μην κοπούν τα κονδύλια για τη συνοχή στο νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και η συζήτηση αυτή νομίζω ότι προσθέτει επιχειρήματα προς την πλευρά που ως Επιτροπή υποστηρίζουμε. Ότι η πολιτική συνοχής δεν πρέπει να θυγεί, πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική, αλλά όχι με περικοπές κονδυλίων. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you. Σας ευχαριστούμε κύριε Παπαδημούλη. Θα έχουμε την ευκαιρία να ε, ε καλέσουμε και κάπως υπουργού από κράτη-μέλη για να λάβω μέρος στη συζήτηση ε, της ε, Επιτροπής. Το είχαμε πει και στις αρχές του μήνα. Συνεχίζουμε με τους υπόλοιπους ε, σκιώδης Η κυρία Ρέντκε απουσιάζει, ε, την αναπληρώνει κάποιος. Όχι, η κυρία Νταμάτο τότε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση του συναδέλφου Αριμών αξιολογεί τα ειδικά μέτρα που εγκρίναμε εμείς το 2015. Την αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης στο 100% και μια προχρηματοδότηση επιπρόσθετη για 7% στα επιχειρησιακά προγράμματα. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τον εισηγητή όταν εύχεται να έχουμε περισσότερα στοιχεία όχι μόνο για το ποσοστό απορρόφησης αλλά και για την ποιοτική εξέλιξη, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και το κοινωνικό ε, όφελος των έργων. Όμως τον Απρίλιο είδαμε ότι η κατάσταση της Ελλάδας μπορεί ακόμα να θεωρείται ειδική λόγω των ε, αδυσβάσταχτων μέτρων που επιβλήθηκαν και του κοινωνικού κόστους που έχει ε, επομιστεί η Ελλάδα εξαιτία της Τρόικας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε εάν τα δημόσια κονδύλια των Ευρωπαίων φορολογουμένων ε, δαπανώνται σωστά και αν έχουν αποφύγει την κατασπατάληση. Θα πρέπει να σκεφτούμε τα ειδικά μέτρα ε, ότι χρησιμεύουν, χρησιμεύουν, όπως ε, το αναφέρει και η έκθεση, σε αυτήν την ε, χώρα με ιδιαίτερες ανάγκες που έχει πολύ μεγάλη ευπάθεια αυτή τη στιγμή λόγω της, των πληγμάτων που έχει δεχτεί ο κοινωνικός της ιστός και η οικονομία της. Θέλω λοιπόν να απευθύνω έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ελπίζω ότι είναι εδώ και θα μας πει και κάτι σχετικά και προς τους συναδέλφους σε ό,τι αφορά το πακέτο νέων κανονισμών. Σίγουρα όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να προσπιστούμε την πολιτική συνοχή που συνεχίζει να είναι η μόνη πολιτική η οποία πραγματικά να διανέμει το εισόδημα και πρέπει να επαγρυπνήσουμε ώστε πέραν του ΑΕΠ όπως έχει υποσχεθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υπάρχουν και άλλοι δείκτες που λαμβάνονται υπόψη όπως η ανεργία των νέων δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα, όπως και η Ιταλία, ιδίω ο νότος της Ιταλίας, έχει πληρώσει το τίμημα, το υψηλότατο τίμημα για την οικονομική κρίση, αλλά και την γενεοδορία την γενεοδορία της, την πραγματική και το υπογραμμίζω, ουσιαστική αλληλεγγύη προς τους ε, μετανάστες σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό λοιπόν και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη δική μας πρόταση που θα προκύψει από το έργο μας εδώ για το ε, επόμενο πλαίσιο 2021-2027 δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν στην πράξη κάποιες αντιφάσεις σε σχέση με τις πολύρες αναγγελίες και τα ωραία λόγια που ακουγόνται πολλές ε, φορές και από το ίδιο το Κοινοβούλιο στις τοποθετήσει του. Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε τα σχόλια των σχεδόν συγκεκριτών. Η κυρία Σπυράκη τώρα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον κύριο Πασκάλα Ριμόντ για την έκθεσή του και να επιβεβαιώσω ότι μετά από μακρύ δρόμο τελικά φτάσαμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα παρά το γεγονός ότι θα ήταν επιθυμητό η έκθεση αυτή να έφτανε στην αρμόδια επιτροπή τη χρονική στιγμή που η Ελλάδα χρειαζόταν ένα θετικό σημάδι. Παρ' όλα αυτά το αποτέλεσμα της έκθεσης είναι ήδη καλό, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι θα επιμείνω σε κάποιες λεπτομέρειες, τις οποίες θα κάνω και τροπολογίες, γιατί πιστεύω ότι καμιά φορά ο διάβολος περιμένει και κρύβεται στις λεπτομέρειες. Πρώτα απ' όλα θεωρώ σημαντική την έλλειψη ότι δεν αναφέρονται στο κείμενο της έκθεσης οι συνθήκες υπό τις οποίες ενεργοποιήθηκε η εξαίρεση, ο κανονισμός 2015-1839 για την Ελλάδα, ο οποίο προέβλεπε και την αύξηση τη προχρηματοδότηση τη τρέχουσα προγραμματική περίοδου τη πολιτική συνοχή και την αύξηση των μεγίστων ποσοστών συγχρηματοδότηση στο 100% για το ανώτατο όριο πληρωμών για την περίοδο 2007-2013. Είναι λοιπόν απαραίτητο να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο με βάση το οποίο θα δίνουμε την εξαίρεση. Διότι μπορεί να θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο δώσαμε στην Ελλάδα την ευκαιρία να μπορέσει να ολοκληρώσει έργα της προηγούμενης περίοδου και να προχωρήσει στη χειρότερη στιγμή τη, όμως η κρίση είναι πάντοτε εδώ. Ως εκ τούτου η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο έχει μια τεχνογνωσία απέναντι σε αυτό το θέμα. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε τα δεδομένα. Και τα δεδομένα που δόθηκαν στην Ελλάδα αυτή την εξαίρεση είναι η Ελλάδα έχασε το 26% του ΑΕΠ της την περίοδο της κρίσης. Η ανεργία εκτινάχτηκε. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχει στη διάθεση της Eurostat το Νοέμβριο του 2017 η Ελλάδα έχει ανεργία 20,9% ενώ η ανεργία στους νέους είναι στο 43,7%. Και αυτά είναι δείκτες και στοιχεία που πρέπει να μείνουν στη συλλογική μνήμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν ενεργοποιεί τέτοιου είδους εξαιρέσεις. Το δεύτερο στοιχείο αυτής της έκθεσης αφορά στην επιμονή της ύπαρξης δικτών ποιοτικού αποτελέσματος. Για όλους μας οι δείκτες ποιοτικού αποτελέσματος παραμένουν το ζητούμενο. Είναι όμως κατά τη γνώμη μου άστοχη η επιμονή να ζητήσουμε από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή να εμφανίσει αυτή μόνη ως κράτος μέλος δείκτης ποιοτικού αποτελέσματος. Και είναι περισσότερο άστοχη η ενέργεια να επιμείνουμε για να δοθεί περαιτέρω και μεγαλύτερη δημοσιότητα για τα έργα που ολοκληρώθηκαν βάσει της εξαίρεσης του 2015. Οι κανόνες δημοσιότητας των συγχρηματοδοτούμενων έργων, οι ταμπέλες που στείλουμε στα συγχρηματοδοτούμενα έργα είναι οι ίδιοι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν χρειάζεται κάτι επιπλέον να κάνει η Ελλάδα σε αυτό. Το τρίτο που θα ήθελα να πω αφορά στην αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Εκεί θα ήθελα να αρκεστώ στο βασικό συμπέρασμα που έβγαλε η Task Force για την Ελλάδα, στο οποίο αναφέρεται ότι για να βελτιωθεί η παροχή της τεχνικής βοήθειας στην Ελλάδα χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα. Θα ήθελα εδώ να μου επιτρέψετε να σημειώσω το εξής. Αυτή η έκθεση για μένα αποτελεί την ευκαιρία για την έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στο πνεύμα της εξαίρεσης που δόθηκε στην πατρίδα μου τον Οκτώβριο του 2015. Ήμασταν εδώ όλοι όταν ζητήσαμε και υπερψηφίσαμε την διαδικασία της άμεσης αλλαγής του κανονισμού. Όμως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο πώς επικοινωνούμε σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. Αυτή η εξαίρεση είναι η έκφραση της αλληλεγγύης. Δεν είναι η ευκαιρία για την αναπαραγωγή στερεοτύπων. Είναι λοιπόν ανάγκη μέσα από όλο το πνεύμα της έκθεσης αλλά και από τις λεπτομέρειές της να επιβεβαιώσουμε τις προσπάθειες του ελληνικού λαού και να αποφύγουμε οποιαδήποτε υπόνοια ότι τα κοινοτικά κονδύλια δόθηκαν με τη μορφή ελεημοσύνης. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Papadakis. Ευχαριστώ κύριε Παπαδάκης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το ομολογείται μέσα στην έκθεση ότι τα κονδύλια δίνονται από το 2011 με τη συνοδεία ειδική ομάδα εργασία για τη στήριξη των λεγόμενων μεταρρυθμίσεων. Δηλαδή πιο συστηματοποιημένα σε σχέση με το παρελθόν, λέγοντα μεταρρυθμίσει, εννοείται και προωθείται όλα τα αντεργατικά μέτρα και τους αντιδραστικούς μηχανισμούς εδραίωσής του που καταρρυπά εξαπολύει ε, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι προηγούμενες αλλά και η σημερινή κυβέρνηση Ριζανέλ στην Ελλάδα σε βάρος των εργαζομένων, των φτωχών απασχολουμένων της μικρομεσαίας αγροτιάς. Επειδή αναφέρεται εδώ για έργα, για μεγάλους εθνικούς δρόμους, θα σας φέρουμε ένα παράδειγμα τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στην βόρεια, στα βόρεια της χώρας, στην Καβάλα, που γίνονται μεγάλες κινητοποίησεις σήμερα οργανώνονται, ακριβώς γιατί στην Εγνατία Οδό από πέρσι επιβάλλονται 13 νέα διόδια τα οποία πληρώνουν πάλι αυτοί που πληρώσαν, γιατί, τα, γιατί οι εθνικοί οδοί κατασκευάζονται με χρήματα των εργαζομένων. Πληρώνουν λοιπόν διόδια διαρκώς περισσότερα, διαρκώς πιο ακριβά και βεβαίως οι κάτοικοι ε, διαμαρτύρονται γιατί εκτός των άλλων ε, προκειμένου να υπάρξει παράκαμψη των διοδίων των καινούριων που μπαίνουν στην Εκνατία Οδό αναγκάζονται να μπαίνουν μέσα από την πόλη της Καβάλας επιβαρύνοντας και περιβαλλοντικά ε, και κυκλοφοριακά την πόλη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της αντεργατικής πολιτικής, της κατασκευής δρόμων προς τα συμφέροντα των μεγαλοκατασκευαστών που οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να τους ε, διανύσουν και πηγαίνουν από τον παράδρομο. Γιατί είναι πανάκριβα παρότι οι ίδιοι τα πληρώσαν. Αυτά είναι αυτή είναι η ποιοτική αξιολόγηση και η κατεύθυνση ε, των έργων αυτών της, ε, που ε, κατασκευάζονται όλα αυτά τα χρόνια. Τα ρεκό λοιπόν της, απορο... της απορροφητικότητας αυτών των κονδυλίων αποδείχθηκε ότι δεν έχουν αποδέχτη το λαό, έχουν τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό ε, αποτυπώνεται και στην έκθεση που λέει για 63% του συνόλου των πληρωμών είναι προσέργα κρατικών ενισχύσεων που αφορούν ενισχύσεις για επιχειρήσεις και επιχειρηματικά σχέδια και το υπόλοιπο 37% αφορά δράσεις κρατικών ενισχύσεων για έργα υποδομών συμπληρώνοντας όπως λέτε τις ρυθμίσεις στον τομέα των συνθηκών της αγοράς και της βελτίωσης των επιχειρήσεων. Δηλαδή μονάζιγα όλα για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Να λοιπόν γιατί τα ευρωνοσιακά κονδύλια και τα κονδύλια των κρατών μελών είναι πλούτος που ανήκει στους εργαζόμενους, αυτοί τον δημιούργησαν και αυτοί πρέπει να τον διεκδικήσουν από όσου τον ληστεύουν τα μονοπόλια, τις αστικές κυβερνήσεις και τις ενώσεις τους. Thank you. Σας ευχαριστώ. δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο από την ομίγυρη, να τον δώσω στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Νέισλερ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη συγγετά και αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ρέγκη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων. να απολύσουμε την κατάσταση κατά το δεύτερο εξάμεινο του 2015, όπου το ελληνικό κράτος και οι ελληνικές τράπεζες αντιμετώπισαν τεράστια προβλήματα ρευστότητας. Ήταν σαφές για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και για όσους χειριζόμαστε τα διαρθρωτικά ταμεία ότι αντιμετώπιζαμε σοβαρό κίνδυνο όλη η εφαρμογή να αποτελματωθεί να κολλήσει και επίσης είχαμε επίγνωση ότι μια τέτοια κινητοποίηση θα είχε σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο και θα επιδίνωνε την κρίση που ήδη ε, σοβούσε. Οπότε ήταν απαραίτητη μια αντίδραση στην κατάσταση, απλή, τολμηρή. Ε, από την άποψη ότι κινητοποίησε ε, πολύ σημαντικά ποσά και μάλιστα άμεση εφαρμογή. Αυτά ήταν τα τρία μέτρα που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την τροποποίηση του κανονισμού των, ε, των κοινών διατάξεων. Δηλαδή, αύξηση τη χρηματοδότηση στο 100% με ένα χρονικό περιορισμό το, ε, για τις ενδιάμεσες πληρωμές στην άρση του ανώτου του ορίου το 95% και επιπλέον 7% προκαταβολές για τη νέα περίοδο 2014-2020. Επίσης να προσθέσω κάτι που ήταν πολύ σημαντικό σε ασφαλιστική δικλίδα. Δηλαδή υπήρχε υποχρέωση του ελληνικού κράτους να δρομολογήσει όλα τα κονδύλια και όλες τις συναφείς πληρωμές μέσω ενός συγκεκριμένου ε, ξεχωριστού λογαριασμού που θα χρησιμοποιούνταν απλώ για τι πληρωμές στους δικαιούχου. ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι οι πληρωμές θα φτάσουν, τα κονδύλια θα φτάσουν στου δικαιούχου σε αυτού που εφάρμοζαν πραγματικά αυτά τα προγράμματα. Έτσι, το 2017 με 2013 πληρώσαμε μία μονοκοντιλιά περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ μέσω της χρηματοδότησης και για το ε, περίοδο μέχρι το 2020 εξασφαλίσαμε την άμεση ε, ταχεία μάλλον ε, έναρξη των προγραμμάτων για τη νέα περίοδο προγραμματισμού. Τώρα εξετάζοντας την αξιολόγηση που στηρίζεται στις, στα στοιχεία που μας έδωσε η ελληνική κυβέρνηση και την έκθεση της ε, τελικές εκθέσεις εφαρμογής που λάβαμε από την Ελλάδα μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι και στις δύο περιπτώσεις τα μέτρα εφαρμόστηκαν επιτυχώς. Για τα προγράμματα του 2007-2013 είχαμε άμεσες ε, παροχές κεφαλαίου κατά το 2015 και οι επιπλέον προκαταβολές εξασφάλισαν άλλες μεταφορές κονδυλίων ε, ενός δισεκατομμυρίου για το 2015 και 2016. Μέσω αυτών των ε, ενέσεων ρευστότητας η Ελλάδα ε, έφτασε σε απορρόφηση 100% των διαθέσιμων κονδυλίων για την περίοδο 2007-2013. Σε σχέση με το μέσο όρο απορρόφησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήταν γύρω στο 96%, η Ελλάδα με 100% ήταν η πρώτη χώρα ως προς την απορρόφηση. Επίσης, τα κοινοτικά κονδύλια έφταναν στην Ελλάδα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Τώρα, στη διαδικασία του κλεισίματος των λογαριασμών, αυτή βαίνει καλώς, εύρυθμα, τακτικά και με βάση τα στοιχεία που έχουμε λάβει μέχρι στιγμή, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν θα έχουμε καμία απώλεια κονδύλιων για την Ελλάδα. Ο αριθμός των τελών προγραμμάτων έχει μειωθεί δραστικά και σε σύγκριση με την περίοδο 2000-2006 και είχαμε 900 σχέδια που δεν ολοκληρώθηκαν. Ενώ στην περίοδο αυτή, 2007-2013, μόνο 79 σχέδια παρέμειναν ατελή. Αν ολοκλήρωτα και που θα ολοκληρωθούν με τη χρήση των εθνικών κονδυλίων. Χωρίς όμως αυτά τα ειδικά μέτρα αυτός ο αριθμός των ανολοκλήρωτων προγραμμάτων θα ήταν ε, πολύ πιο μεγάλος και η Ελλάδα θα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα κονδύλια και, να, και για να ολοκληρώσει αυτά τα σχέδια και προγράμματα. Η Ελλάδα κατάφερε επίσης να ολοκληρώσει πολύ σημαντικά σχέδια και προγράμματα. Ο κύριος Αριμόν ανέφερε τα πιο εμβληματικά ε, οι παραχωρήσεις για τους αυτοκινητοδρόμους, για παράδειγμα. Ήταν πολύ σημαντική επιτυχία. Και έτσι μπόρεσαν να συνεχιστούν τα έργα και το 2017 και τα πέντε προγράμματα, σχέδια μάλλον, ε, ολοκληρώθηκαν και εγγενιάστηκαν. Και χάρη στην ε, έκτακτη 7% εμπροστοβαρή ε, χρηματοδότηση για, το, για την περίοδο μέχρι το 2020. Η απορρόφηση ε, για την περίοδο αυτή έχει φτάσει μέχρι το 25% και ενώ 14% είναι ο κυρωτικό μέσο όρο. Ακόμη και αν αποκλείσουμε την αύξηση του 7% τη προκαταβολή, τη επιπλέον προκαταβολή, ακόμη και χωρί αυτό, η Ελλάδα έχει πολύ καλύτερε επιδόσει από τον κοινοτικό όρο ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι η Ελλάδα υποχρεώθηκε να δικαιολογήσει αυτή την ε, αύξηση της προκαταβολής του 7% υποβάλλοντας κάποιες ε, ενδιάμεσες ε, διεκδικήσεις πληρωμών που διεκπαιρεώθηκαν αισίως. Τώρα βλέπουμε ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει σε μια σωστή πορεία σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των διαρθρωτικών κονδυλίων και είναι από τις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις στον τομέα αυτό. Να προσθέσω και λίγα λόγια γιατί πολλά μέλη της Επιτροπής αναφέρθηκαν στο ζήτημα της ανταγωνιστικότητας. Η κατάσταση είναι τέτοια που δεν είχαμε την υποχρέωση να αξιολογήσουμε πόσο ο συνολικός αντίκτυπος ε, των μέτρων επηρέασε τις μακροπρόθεσμες προοπτικές. Αυτό θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο του κατά πόσο τα μέτρα ε, εφαρμόστηκαν επιτυχώς στο συγκεκριμένο πλαίσιο και η απάντηση είναι ανεπιφύλακτα καταφατική. Ε, τώρα στο θέμα της ανταγωνιστικότητας ε, το θέμα αυτό θα πρέπει να το δούμε με πιο μακροπρόθεσμη προοπτική και εκεί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και κάποιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που συνεχίζονται στην Ελλάδα και που οπωσδήποτε θα πρέπει να αξιολογηθούν ε, πιο διεξοδικά. Πάντως από μέχρι τώρα εκθέσεις ε, από τις πηγές της Παγκόσμιας Τράπεζας αλλά και από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα έχει αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της σε σχέση με πριν από μία πενταετία. Οπότε η συνολική εκτίμηση και το γενικό συμπέρασμα είναι πολύ θετικά. Και να είστε βέβαιοι ότι η συμβολή, η συνεισφορά των διαρθρωτικών ταμείων στην ε, γενική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας ε, ε, τη χάνει μόνιμης αξιολόγησης στα πλαίσια και του μνημονίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Αριμό για την άρτια έκθεσή του και για την πολύ ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων που είχαμε και με τους συναδέλφους και με το επιτελείο, το προσωπικό γραφείο της Επιτρόπου Κρέτσου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αρημό, Για να ολοκληρώσουμε. Ναι, δεν θα ήθελα να πω πολλά πράγματα. Νομίζω ότι όλα έχουν υποθεί όσα πρέπει να υποθούν. Χαίρομαι για την συνεργασία με τους συναδέλφους προκειμένου να ολοκληρωθεί και να βελτιωθεί αυτή η έκθεση. Το χρονοδιάγραμμα και η ημερομηνία κατά την οποία, μέχρι την οποία θα πρέπει να υποβληθούν τροπολογίες ε, είναι σύντομο. Θα πρέπει λοιπόν να βιαστούμε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επιτροπή για την καλή συνεργασία που είχαμε. Στο τέλος της ημέρας, ε, όχι τελικά, συγγνώμη, θα ολοκληρωθεί η έκθεση αυτή. Ε, και θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε ότι η περιφερική πολιτική και υπό δυσχερείς ε, συγκυρίες είναι το δεδειγμένο εργαλείο για να στηριχθούν χώρες που βρίσκονται σε δυσκολίες και νομίζω ότι μπορεί με τον τρόπο αυτό να προβληθεί και η περίπτωση της ε, Ελλάδος ως ε, πετυχημένο παράδειγμα υποδοχής ειδικών μέτρων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η προθεσμία υποβολής των τροπολογιών είναι 6 το απόγευμα, 7 Μαΐου, στις 17 Μαΐου, συγγνώμη, ε, πράγματι είναι σε... πολύ σύντομα. Ε, είδατε ότι ήταν θετική η υποδοχή της έκθεσής σας, άρα μάλλον θα είναι περισσότερο ο αριθμός των τροπολογιών, αλλά εν πάση περιπτώσει η κοινή θέση της Επιτροπής είναι ότι πρόκειται για μια πολύ καλή έκθεση. 17 Μαΐου, 6 το απόγευμα, ε, προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών και θα ψηφιστεί η έκθεση κατά τη συνεδρίασή μας του Ιουνίου αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπερψηφιστεί ούτε ώστε να αποτελέσει ένα θετικό μήνυμα όσον αφορά την υποδοχή των ειδικών μέτρων που έλαβε η Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας ε, διάταξης. Είναι η παρουσίαση της μελέτης νέες τεχνολογίες και περιφερειακή πολιτική στο, νέο, στο, πλαίσιο, στο νέο πλαίσιο ε, πολιτικής ε, συναχής ε, έχει γίνει ένα εργαστήριο και στη συνέχεια εκπονήθηκε μία έκθεση η οποία συζητήθηκε στο πάνελ ε, της ΣΤΟΑ στις 8 Φεβρουαρίου και τώρα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την παρουσίαση αυτής της έκθεσης για τις νέες τεχνολογίες και περιφερειακή πολιτική και έχω τη χαρά να καλέσω τον καθηγητή κύριο Άνερστετ να μας παρουσιάσει την ε, μελέτη αυτή. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους. Ε, έχω 15 λεπτά για να σας πείσω ότι η έκθεση αυτή των 69 σελίδων αξίζει να διαφαστεί, τουλάχιστον να την ξεφυλίσετε. Έχετε επίσης τέσσερις σελίδες σύνοψης που περιλαμβάνουν δέκα συμπεράσματα. Νέες τεχνολογίες προς ένα νέο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Όπως είπατε, έγινε ένα εργαστήριο τον προηγούμενο Οκτώβριο και εγώ το πήρα πολύ σοβαρά, όχι μόνο για να συνοψίσω το τι περιέλαβε, αλλά προκειμένου να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες για την ε, περιφερειακή ε, πολιτική όσον αφορά την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και την πολιτική συνοχή επιφέροντας τις, ε, προσθέτοντας τις διαστάσεις της, των καινοτομιών. Και πραγματικά χάρηκα που άκουσα τις δικές απόψεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνεται λοιπόν από αυτό το workshop και αυτή η σάθος έκθεση ε, αναφέρει ότι οι ψηφιακές οικονομίες και νέες τεχνολογίες είναι ένα κατάλληλο εργαλείο για την ενδυνάμωση της πολιτικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εξετάσω ορισμένες πτυχές που προωθούν αυτή την ε, μεταφορά από την ε, ψηφιακή τεχνολογία στην ε, παραγωγή. Άρα λοιπόν αφορά πάρα πολύ τα όσα συζητείτε εδώ στο πλαίσιο των εκθέσεων και με τις προσεχείς μήνες όσον αφορά το μέλλον του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Οι εισφορές στο workshop δόθηκαν από την Κομισιόν και τις χώρες μέλη. Ήταν μια σειρά από δραστηριότητες ε, παρακολούθησης και διάφορες ε, αξιολογήσεις των πολιτικών που μου διαφυβάστηκαν και επίσης και υπήρξε και επιστημονική έρευνα. Ε, αυτό ήταν το, το πλαίσιο της έκθεσης. Όπως σας είπα, περιλαμβάνει 69 σελίδες η μελέτη αυτή ε, και βεβαίως θα δεχτώ, ε, είμαι πρόθυμος να δεχτώ και τις, ε, τα δικά σας σχόλια και να τα προσθέσω, να συμπεριλάβω. Το... Υπάρχει μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών μεγάλες αποκλίσεις. Αυτή είναι η το σημείο εκκίνησης. Υπάρχουν περιφέρειες οι οποίε δεν εξελίσσονται ταχαίω. Ένα από τα σημεία που αναφέραμε στην ε, μελέτη είναι ότι κάθε περιφέρεια έχει διακριτά χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει μια πανάκια, μια συνταγή για όλες τις περιφέρειες. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Άρα θα πρέπει να υπάρξει ένα ε, μια μεγάλη ευελιξία και αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο της μελέτης αυτής. Θα πρέπει να εξάβρουμε την ευελιξία, τη διαδικασία fast track κλπ. ούτε ώστε η κάθε μια από τις περιφέρειες να μπορεί να αξιοποιήσει τα κονδύλια τα οποία και τεχνική συνδρομή που λαμβάνει εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βασική έννοια ε, είναι το πώς η τεχνολογία δυναμώνει την παραγωγικότητα και, την, ε, και πώς, οι, πώς αξιοποιούνται οι καινοτομίε. Η Ευρώπη είναι στην πρώτη θέση όσον αφορά τις ε, τεχνολογίες επικοινωνίες. Η Γερμανία οι Γερμανοί και οι Βρετανοί ε, ειδικοί είναι αυτοί οι οποίοι κατασκεύασαν τους πρώτους υπολογιστές και προώθησαν όλη την ε, ψηφιακή τεχνολογία, αλλά δεν μπορέσαν να εξοπλίσουν αυτό το κεφάλαιο. Η περαιτέρω εξελίξη έγιναν από τους Αμερικανούς, Κινέζους κλπ. Άρα λοιπόν η Ευρώπη διαθέτει ένα τεράστιο επιστημονικό δυναμικό όσον αφορά τι ε, τεχνολογικέ επινοήσει, αλλά, δεν, αλλά όσον αφορά το, τη μεταφορά. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν προς τα πού πηγαίνει η ευρωπαϊκή προστάμενη αξία. Μπορούμε να βελτιώσουμε περαιτέρω το τεχνολογικό μας δυναμικό και να το μεταφέρουμε στην οικονομία της κάθε περιφέρειας. Ε, αυτό είναι το θέμα. Άρα τα θέματα κλειδί, έτσι όπως τα βλέπω, είναι του πώς ε, μπορεί να γίνει αυτή, αυτό το transfer, αυτή η μεταφορά στο επίπεδο της οικονομίας. Ε, η καινοτομία στα πέτα της ε, αριστείας είναι το πρώτο στοιχείο. Η αξιοποίηση της ε, έξυπνης εξειδίκευσης αλλά εστιάζοντας στην πολιτική αντικτύπου. Ε, θεωρώ ότι αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο. Πρόκειται για μια πολύ καλή άσκηση, η οποία εφαρμόζεται στο επίπεδο πολλών περιφερειών και οδηγεί στην, ε, σε μια μορφή συνεργασίας μεταξύ πολιτικής και επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Δεν λέω ότι κάθε περιφέρεια θα πρέπει να στείλει κάποιο στο φεγγάρι, αλλά αναφέρομαι στην διατύπωση κοινωνικών και οικονομικών στόχων στο επίπεδο της κάθε περιφέρειας, ώστε να δούμε τι γίνεται με την προώθηση μιας έξυπνης εξειδίκευσης στο επίπεδο των περιφερειών. Εάν δούμε τις ε, προτάσεις της Επιτροπής, ε, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση ε, στο, στην ενεργοποίηση των περιφερειακών αρχών στους τομείς αυτούς. Και θα πρέπει να θυμηθούμε μια έννοια κλειδί ε, να έχουμε κατά νου μάλλον μια έννοια κλειδί, είναι η δυναμική τοποθέτηση. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Είναι το να σκεφτούμε περισσότερο και πιο γρήγορα, ε, πιο ενεργές ε, πολιτικές δράσεις. Εάν έχουμε μια κατευθύνση σε ένα κοινωνικό και οικονομικό στόχο, θα πρέπει να διατυπωθεί και να προβληθεί προς τον κοινό προς το τομέα της, ε, για να προβληθεί στην κοινή γνώμη, ώστε να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ των διαφέρων ε, φορέων και αυτό θα οδηγήσει σε μια νέα, ένα, πολιτική marketing ε, και συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αξιοποιώντα τι πιο πρόσφατε ψηφιακέ, όχι μόνο ψηφιακέ τεχνολογίε, αλλά και άλλε τεχνολογίε, διαμορφώνοντα ε, μια νέα μορφή marketing. Για να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο τη περιφερειακή πολιτική, πολλέ από αυτέ δεν συνδέονται με τις ε, παγκόσμιες μεταβολές και βλέπουμε ότι ορισμένε περιφέρειες είναι πετυχημένες αυτές του νέου τύπου marketing. Για παράδειγμα, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία η οποία έκανε μια επανάσταση στο επίπεδο μιας υπάρχουσας υποδομής δημιουργώντας, κάνοντας ε, δημιουργώντα ταχύε εξελίξει όχι μόνο στον τομέα αυτό τη αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά έχοντα θετικά αποτελέσματα και στου άλλου βιομηχανικού τομεί. Η η οικονομία της, των ψηφια, της ψηφιακής πλατφόρμας είναι σημαντική. Αν μιλούμε για τεχνολογία σήμερα και δούμε τι γίνεται πριν από 10 χρόνια, πρόκειται για μια επανάσταση το πώς η τεχνολογία αξιοποιείται στο επίπεδο της περιφερειακής ε, ανάπτυξης. Ε, και θα πρέπει να υποτιμούμε ε, το τομέα αυτό. Εμείς συνεισφέραμε πολύ όσον αφορά την ανάπτυξη αυτών των, ε, της ψηφιακής, ε, ε, στις ψηφιακές πλατφόρμες στη Δανία και σε άλλες χώρες αλλά είναι Αμερικανοί και πάλι αυτοί οι οποίοι προώθησαν περαιτέρω αυτές τις καινοτομίες. Και τώρα εμείς στην Ευρώπη αρχίζουμε να εφαρμόζουμε αυτά τα οποία οι Αμερικανοί έκαναν ε, στο παρελθόν. Τέλος, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στο επίπεδο του ενός καινοτόμου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν, αυτές οι υποδείξεις έτσι όπως τις έχετε ε, στη σύνοψη των τεσσάρων σελίδων μπορείτε να ανατρέξετε τις συστάσεις. Θα ήθελα να τονίσω τα εξή όσον αφορά την οικονομία στις ψηφιακές πλατφόρμες. Είναι πολύ σημαντικό οι περιφέρειες να δουν τις εναλλακτικέ δυνατότητες και τις ευκαιρίες του μάρκετινγκ της διασύνδεσης με τους ε, βασικούς ε, πελάτες ακόμα και σε ε, περιορισμένες αγοράς γιατί εάν αθρηστούν ε, μπορούν να αποκτήσουν καθοριστική σημασία προκειμένου και οι απόμακρες περιοχές της Ευρώπης να μπορέσουν να έχουν μια πρόσβαση σε μια πελατεία. Όσον αφορά την ψηφιοποίηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ ενεργό ρόλο και είναι πολύ έξυπνη όσον αφορά την ψηφιοποίηση. Έχουμε τα digital hubs, τους ψηφιακούς κόμβους, οι οποίοι μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους ε, καλύτερα, να υπάρξει πιο στενή συνεργασία με το ιδιωτικό τομέα κλπ. Επίσης τα λεγόμενα science parks, τα πάρκα επιστήμης, αλλά και άλλες ε, καινοτομίες και επαγγελματική διαχείριση όλων αυτών των καινοτόμων ε, τομέων. Δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε τις αλλαγές κοινότητε που υπάρχουν στο επίπεδο των περιφερειών όσο εξάρτητα από το κατά πόσο προθυμένες τεχνολογικά είναι οι περιφέρειες αυτές και έχουμε αυτές τις συνεργασίες με κεφάλαια ψηλού επιχειρηματικού κενδύνου, με πανεπιστήμια κλπ. Ε, πρόκειται για αναλυτικέ δυνατότητες οι οποίες θα έπρεπε να ληφθούν πολύ σοβαρά. Τώρα, η δική μου πρόταση ε, είναι ακριβώς αυτή η έννοια του dynamic positioning, της δυναμικής τοποθέτησης. Χρειαζόμαστε άμεσες κάθετες πολιτικές. Χρειάζεται καλύτερη διαχείριση των διαδικασιών fast track. Πολλές φορές ε, μου είπαν ότι τέτοιες ταχείες δράσεις είναι αναγκαίες για να καλύψουμε τα κενά της ε, βραδίας ε, διαδικασίας και να τις μετατρέψουμε σε πιο αποτελεσματικές πολιτικές, δεσμεύοντας επίσης και τον ιδιωτικό τομέα και προωθώντας με ένα πιο ενεργητικό τρόπο τις διαδικασίες fast track, οι οποίες ε, μπορούν να προωθήσουν την συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ε, δεν θα πρέπει να αναμένουμε αυτές τις διαδικασίες, αλλά θα πρέπει να προωθήσουμε ε, περισσότερες ε, καινοτομίες ταχύτερα. Αυτό είναι σημαντικό για την πολιτική συνοχής προκειμένου να προχωρήσει στο προσεχές δημοσιονομικό πλαίσιο και είναι σημαντικό να έχουμε μία ε, ταχεία εξέλιξη προκειμένου να γίνουν ε, αποτελεσματικά οι αναγκαίες επενδύσεις. Τι σημαίνει αυτό συγκεκριμένα. Θα πρέπει να γίνεται μια σωστή οικονομική εκτίμηση στο επίπεδο της κάθε περιφέρειας και να πρέπει να θαρρύνουμε τις περιφέρειες να αναλάβουν πιο ενεργητικό ρόλο, να μην αναμένουν, ε, παθητικά την εφαρμογή των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, αλλά να λειτουργούν σε μια συνεχή βάση ε, ως μια συνεχιζόμενη διαδικασία και όχι μια διαδικασία ε, σε δύο ή τρεις φάσεις. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να υπάρχει μια ευέλικτη πολιτική καθοδήγηση και αυτό φορά και την Επιτροπή και την Οικονομική Ένωση. Θα πρέπει να προβληματιστεί σε σχέση με την ευελιξία η οποία παρέχεται και με τον, την ε, ε, εφαρμογή, τη ε, αυτών των πολιτικών και πρέπει, θα πρέπει να υπάρχει ένα συνεκτικό, μια συνεκτική δέσμη δράσεων γιατί η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία και ο υπόλοιπος κόσμος εξελίσσεται πολύ γοργά όπως για παράδειγμα η Κίνα που έχουν αυτές τις διαδικασίες fast track, ε, κατεξοχήν. Ε, και εμείς θα πρέπει να σκεφτούμε με τέτοιους ώρες. Είμαστε πολύ καλοί στην επιστήμη και στην τεχνολογία, αλλά είμαστε λιγότερο καλοί στις καινοτομίες και υστερούμε ακόμα περισσότερο όσον αφορά τις εφαρμογές για τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να κινηθούμε πιο γρήγορα. Τώρα, όσον αφορά την έξυπνη εξεδίκευση, Νομίζω, για μια ευρωπαϊκή επινόηση και δεν είναι μόνο οι επιστήμονες αλλά και οι πολιτικοί οι οποίοι ασχολήθηκαν με αυτό το μοντέλο αλλά θα πρέπει και να εφαρμοστεί. Και αν δείτε την πρόταση που διατυπώνει η Επιτροπή αναφέρεται ότι θα πρέπει να γίνουν κάποια βήματα προς τα μπρος, θα πρέπει να σκεφτούμε εκ νέου το πώς μπορεί να γίνει αυτή η έξυπνη εξειδίκευση. Θα πρέπει να μεταφερθούμε προς μία τζέντα η οποία να στοχεύει στην έξυπνη εφαρμογή. Θα πρέπει να δούμε ποιο ε, θα πρέπει να είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα για την κάθε μία περιφέρεια ε, οι όσον αφορά λυσμένες ε, προσεγγίσεις. Θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα σε αφορά τις επιχειρήσεις, το δημόσιο τομέα, τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων κλπ. Ε, εδώ μπορεί να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Δεν λέω ότι θα πρέπει να... Ε, εγώ λέω ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η έξυπνη εξειδίκευση. Τώρα, ε, υπάρχουν κάποια κρίσιμα θέματα ε, σε σχέση με τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε στρατηγικούς ε, τομείς. Ε, θα πρέπει να υπάρξει μια πιο ενεργητική δέσμευση εκ μέρους των περιφερειακών αρχών όσον αφορά τις μορφές συνεργασίας στον ιδιωτικό τομέα γιατί στα χαρτιά τα πράγματα είναι καλά αλλά όχι πάντα στην πράξη. Μία από τις προτάσεις μου είναι να εμπλέξουμε πιο ενεργά τις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές, να τις εξοπλίσουμε καλύτερα, να τις βοηθήσουμε να αποκτήσουν πιο επαγγελματικό χαρακτήρα, να μπορέσουν να λάβουν κινδύνους, να γίνουν πιο τολμηρές ε, σε ό,τι αφορά τη μέσο και μακροπρόθεσμο, το μέσο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της περιφερειακής ανάπτυξης και να έχουν πιο ενεργές ε, σχέσεις με άλλες περιφέρειες. Η διασυνοριακή συνεργασία έχει μεγάλη σημασία Επίσης, να βοηθήσουμε τους τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες να δουν ξεκάθαρα τη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, να διασυνδεθούν διασυνοριακά, να έχουν διασυνοριακές επενδύσεις σε συνεργασία με τα κράτη και τις περιφέρειες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω κάτι που αναφέρθηκε όχι μόνο στη δική μας έκθεση αλλά και από άλλους ε, φορείς η ανάγκη επενδύσεων προσανατολισμένων ανατολισμένες συγκεκριμένες ε, αποστολές και καθήκοντα. Παράδειγμα η Σουηδία. Είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε πώς οι περιφέρειές μας και οι εταίροι μας αντιμετωπίζουν τις κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις στα θέματα υγειονομικής περίθαλψης, ε, βιωσιμότητας των πόλεων, των δήμων ε, τεχνολογιών, ε, καθαρών τεχνολογιών και ούτω καθεξής. Αν τα δούμε αυτά μαζί με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ε, οργανώσεων ασθενών, μπορούμε να έχουμε ένα πολύ πιο δίκαιο σύστημα καινοτομίας πολύ πιο προορατικό, στρατηγικού σχεδιασμού που θα έχει και αυτά αποτελέσματα για την κοινωνία. Οπότε θα πρέπει να έχουμε επενδύσεις προσανατολισμένες προς τις συγκεκριμένες αποστολές που θα πρέπει να επιτελέσουν και με πιο ενεργό εμπλοκή της κοινωνίας. Έτσι η τεχνολογία και η καινοτομία θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυτή τη διαδικασία. Και πιστεύω ότι από ευρωπαϊκή σκοπιά η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία εδώ θα ήταν τεράστια. Θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις περιφέρειες ε, να σκεφτούν καλύτερα, χρησιμοποιώντας το δανέζικο, το γαλλικό, το σουηδικό παράδειγμα. Έχουμε μία σειρά τέτοιων επενδύσεων προσανατολισμένων προς, τις απο... προς συγκεκριμένες αποστολές που χρησιμοποιήθηκαν ενεργά, προορατικά, με ανάμειξη των περιφερειών ε, και των ε, επιχειρήσεων των περιφερειών που συμπαρατάχθηκαν όλοι σε αυτό το σκοπό. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για να προωθήσουμε καλύτερα την ευφυή εξειδίκευση. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μια δραστηριότητα που διαμορφώνει την αγορά. Οπότε ο δημόσιος τομέας εδώ θα μπορούσε να βοηθήσει. Αυτό συνέβη στις ΗΠΑ, συμβαίνει και στην Κίνα. Σε μεγάλο βαθμό. Η Κινέζικη κυβέρνηση πολύ ενεργά ε, εμπλέκει τον ιδιωτικό κλάδο στη διαμόρφωση των κοινωνικών και οικονομικών προγραμμάτων της και το κάνει η κινέζικη κυβέρνηση πολύ έξυπνα. Και εμείς ε, που είμαστε ένα δημοκρατικό μπλοκ θα πρέπει να το κάνουμε καλύτερα ακόμη γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερες ικανότητες από αυτήν την άποψη από ότι οι Κινέζοι. Και να προσθέσω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Όταν ε, μιλούμε για την περιφερειακή ε, πολιτική και την πολιτική συνοχής δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε αυτόνομα τις περιφέρειες, αλλά τις περιφέρειες ως τμήματα της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν μήπω μήπως οι περιφέρειες δεν έχουν τις, τους πόρους που χρειάζονται για να προσανατολίσουν σε επενδύσεις τους σε αποστολές. Οπότε θα πρέπει να τις βοηθήσουμε να βρουν εταίρους και εκτός του πλαισίου τους. Και μάλιστα αυτό θα πρέπει να το κάνουμε πιο συστηματικά ε, αναλύοντας τα παραδείγματα που σας προανέφερα. Στη Σλοβακία, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να αναβαθμίσουμε ολόκληρο κλάδο και να τον φέρουμε στην πρωτοκαθεδρία, επηρεάζοντας και άλλους τομείς. Και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε μόνο με μια καλύτερη διασύνδεση των σλοβακικών περιοχών με άλλες εκτός της Σλοβακίας περιφέρειες. Αυτά ήταν μερικά από τα σημεία που πραγματεύεται η έκθεση που όπως σας είπα έχει 69 σελίδες. Ελπίζω να σας έδωσα τροφή για σκέψη και να σας ξύπνησα το ενδιαφέρον για να διαβάσετε αυτή την έκθεση. Νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ ε, σημαντική στιγμή, πολύ κρίσιμη στιγμή και πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή της πολιτικής και μια επιτροπή σε τη δική σας, ε, άνθρωποι σαν και εσάς, ε, και ε, οι συνεργάτες σας θα μπορούσατε να προωθήσετε όλα αυτά τα σημεία πολύ πιο δραστηρία και πραγματικά να προτείνετε έλευθες αλλαγές εν ώψη του επόμενου πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή σας την παρουσίαση. Ο λόγο τώρα στον κύριο Βαλκάρσελ Σίσο που είναι ο αρμόδιος αντιπρόεδρος ε, για τη ΣΤΟΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχετε το λόγο κύριε Σίσο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως, έχουμε μία μελέτη που πραγματεύεται ένα πολύ σημαντικό θέμα την ανάπτυξη των ε, τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Ένα ζωτική σημασία ζήτημα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τα ταμεία της συνοχής ήδη χρηματοδοτούν δραστηριότητες ε, εφαρμογής ε, και προγραμματισμού υποδομών τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, η ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων. Η μελέτη ε, περιστρέφεται γύρω από τις ε, πολιτικές συνοχές που βοήθησαν στην ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών, πληροφορίας και επικοινωνίας, μέσω στρατηγικών εφιούς ειδίκευσης, μέσω της ανάπτυξης τέτοιων πάρκων επιστημονικών και τεχνολογικών για να ε, ενισχύσουν την έρευνα και τις ΣΔΙΤ, αλλά προωθώντας και την έρευνα στην ψηφιακή αγορά και στην ανάπτυξη της αγοράς γενικώς. Με τις απαντήσεις που λάβαμε ε, από, μια, από ένα ευρύ φάσμα πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για την μελέτη έχουμε πολύ χρήσιμα στοιχεία. Ε, η μελέτη στηρίχθηκε με στοιχεία των Γενικών Διευθύνσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στοιχεία τη ε, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Επιτροπή των Περιφερειών, αλλά και τη ε, Διεθνού Ένωση Τεχνολογικών Πάρκων από πέντε ευρωπαϊκέ περιφέρειες και πολλά κράτη-μέλη, ενώ ταυτόχρονα ανάλυσε πολύ σημαντικά έγγραφα, όπω είναι η 7η έκθεση τη πολιτική συνοχή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και φυσικά ανέλησε και πολύ περισσότερα έγγραφα και δημοσιεύματα. Νομίζω ότι πολύ λογικά η έκθεση αυτή κάνει μια ανάλυση της παρούσας κατάστασης, περιγράφει την πολιτική πραγματικότητα της πολιτικής συνοχής και της εφίους ειδίκευσης και επισήμανε τις δυσκολίες που εμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση του περιφερειακού δυναμικού με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Η μελέτη αυτή θεωρώ ότι όχι μόνο θα είναι χρήσιμο εργαλείο για να κάνουμε μια επισκόπηση της κατάστασης και των σημείων που χρήζουν βελτίωσης, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μελέτη ως βάση για τις μελλοντικές μας πολιτικές στον τομέα αυτό. Ιδιαίτερα εν ώψη του νέου πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Γιατί με τέτοιου είδου μελέτε μπορούμε να δικαιολογήσουμε την ανάγκη να συνεχίσουμε τι επενδύσει μα στην καινοτομία, στην έρευνα και στα επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα, προκειμένου να έχουμε μια πιο αποδοτική, αποτελεσματική και ανταγωνιστική οικονομία στην Ευρώπη, ε, στο μέλλον που θα έχουμε και μεγαλύτερη σπάνη πόρων. Ευχαριστώ τον κύριο Χόνερστετ για το έργο του στη ΣΤΟΑ και ευχαριστώ και για την παρουσίαση που μας έκανε τις μελέτες αυτής της ΣΤΟΑ. Thank Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κρέλ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, βρήκα πολύ σημαντική την ε, παρουσίαση. Εγώ πρέπει να διαβάσω αυτές τις 65 σελίδες. Έχω όμως ε, έχω την αίσθηση ότι στα συμπεράσματα όσον αφορά την πολιτική συνοχής έχουμε μια εσωτερική σύγκρουση. Λέτε σε πολλά σημεία ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία, πρέπει να υπάρξει πρόσβαση ε, τύπου fast track και ακριβώς, αυτό είναι το οποίο δεν κάνουμε. Δηλαδή τέλη Μαΐου θα πάρουμε τις προτάσεις για το νομικό πλαίσιο Ε, για το 21 έως 28 Δηλαδή τα επόμενα μίση έτος θα αποφασίσουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ε, είναι πολύ αργότερα. Αυτή είναι μια εσωτερική σύγκρουση. Δεν είναι δυνατόν να είμαι ευέλικτο και να αντιδρώ τάχιστα εάν χαράσω, χαράτω μια πολιτική για 7 χρόνια με σταθερούς αλγόριθμους, ε, πάγια στόχευση κλπ. Ε, πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο ε, όσον αφορά το impact focus policy, δηλαδή την ε, πολιτική στόχευση στις επιπτώσεις. Αυτό το συζητούμε εδώ και πολύ καιρό. Πώς θα φύγουμε από την αποκλειστικά οικονομική στήριξη σε έναν προσανατολισμό προς την αποτελεσματικότητα. Εγώ δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Πώς ε, μπορεί να συμπεριληφθεί σε ένα κανονισμό και ποιο θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα. Αναφερθήκατε στην αιρεσιμότητα εξάντε εν συντομία. Αλλά αν ε, σκεφτούμε ότι η Επιτροπή υπαγορεύει μία αιρεσιμότητα εξάντε για την έξυπνη εξειδίκευση, smart specialization. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε εταιρικέ συμφωνίε με τι χώρε μέλη για τα επόμενα χρόνια, τι φαντάζονται. Ε, θα πρέπει να γίνει δηλαδή ε, μια εφαρμογή στο επίπεδο των περιφερειών, ώστε να εκπονηθεί κάποια στρατηγική. Πώς θέλουμε να αναπτύξουμε αυτή την ευελιξία στους τομείς αυτή, πώς ε, θέλουμε να απαντήσουμε στα ζητήματα αυτά τα επόμενα 7 χρόνια μέχρι ότου συγκεντρώσω όλα αυτά τα στοιχεία και ε, να τα διαβάσω πάλι στην Επιτροπή και συζητηθούν όλα αυτά με την Επιτροπή. Θα παρέλθουν άλλα δύο χρόνια. Αλλά τότε αυτό το οποίο είχα αρχικά σαν ιδέα, τότε πλέον θα είναι πεπαλαιωμένο πριν ε, φτάσει η στρατηγική αυτή πάνω στο τραπέζι. Μπορώ να φανταστώ μετά από την επίσκεψή μας στη ΣΥΠΑ όπου το θέμα ήταν και πάλι και καινοτομίε. Μπορώ να φανταστώ γιατί αυτή είναι πιο ευέλικτη. Γιατί δεν έχουν ένα δημόσιο τοπέα ο οποίο ασχολείται με τέτοια θέματα. Έχουν ένα πολύ ευέλικτο τομέα που ο καθένα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει αλλά που δεν υπάρχει μια πρόθεση εκ μέρους των περιφερειών οι οποίες θα πρέπει να χρηματοδοτούν από κάπου αλλού. Εκεί είναι ευέλικτα και είναι όλα ιδιωτικά. Ε, πρόκειται για μια εντελώ, ένα εντελώς διαφορετικό αξιολογικό σύστημα από ό,τι στην Ευρώπη. Γι' αυτό μπορούν να είναι πολύ πιο γρήγοροι από εμά. Κατά πόσο αυτό τελικά είναι καλύτερο, δεν ξέρω. Έχω κάποιες αμφιβολίες γιατί και η Κίνα είναι, στην Κίνα είναι αντίστοιχα τα πράγματα. Ε, κανείς δεν ενδιαφέρεται κατά πόσο υπάρχει ένα δημοκρατικά εκλεγμένο κοινοβούλιο το οποίο κλπ. κλπ. Ε, ε, σκοτούρα τους. Ε, αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν. Ε, και γι' αυτό είναι πιο ευέλικτη και πιο γρήγορη και σε ορισμένου τομεί πιο πετυχημένη. Ωστόσο δεν είναι η πρόσληψη την οποία έχουμε εδώ, το μοντέλο το οποίο ακολουθούμε εδώ στην Ευρώπη. Ε, η δική μας αντίληψη το πώς λειτουργούν τα πράγματα σε μια δημοκρατική κοινωνία ε, εδώ είναι το ζήτημα. Δεν ξέρω, μπορείτε να μου αποδείξετε εσείς κάποια απάντηση. Ευχαριστούμε. Ίσως κάποιος μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις. Ε, κυρία Μάλετιτς, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ καθηγητά για την προσοχή σας, την εξαιρετική αυτή μελέτη. Είναι πραγματικά ύψης της σημασίας να σκεφτούμε ξανά πώς μπορούμε να έχουμε μια νέα προσέγγιση για την πολιτική συνοχής για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα επιτόπου. Η ερώτησή μου είναι ακριβώς για τη θέση της ευφυούς εξειδικεύσης αυτή τη στιγμή στο τωρινό πλαίσιο. Η ευφυής εξειδικεύση ήταν μια ένα εξάντερ κριτήριο ρεσιμότητας για την προτεραιότητα υπαριθμών 1. Δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε έτοιμοι και πόσο έχουμε περάσει στη φάση της ε, υλοποίησης για τη στρατηγική της ευφυούς εξειδικεύσης αυτή τη φάση. Γνωρίζω ότι πολλές περιοχές έχουν προετοιμάσει το έδαφος. Υπάρχουν όμως ε, πραγματικά σωστές καταγραφές των αναγκών. Θα θέλαμε μια νέα έννοια που θα είναι, δεν θέλω να πω πιο περίπλοκη, αλλά αναβαθμισμένη. ώστε να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην πράξη. Χρειάζεται ένας καινούς προσανατολισμός, να επικεντρωθούμε στα αποτελέσματα και όχι στην ε, συνεισφορά μας όχι. Δηλαδή να σκεφτούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τους πόρους μας ε, για σκοπούς ανάπτυξης, να καλύψουμε ανισότητες και διαφορές μεταξύ των ε, περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μπορούμε λοιπόν να πετύχουμε, μάλλον τι νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε για να καταφέρουμε να έχουμε αυτή τη νέα προσέγγιση στην πολιτική συνοχή και να είμαστε και έτοιμοι για το 2021 για να εφαρμόσουμε αυτή τη νέα προσέγγιση στην πολιτική συνοχή. για να μην καταλήξουμε να έχουμε πάλι ένα κριτήριο εξάρτητα ρεσιμότητα που να μπορούμε να το εφαρμόσουμε και πάλι να μπορούμε να το ελέγξουμε και τελικά πάλι να μην έχουμε αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μπρέσο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ τον καθηγητή για την ε, ε, έκθεση αυτή που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ήθελα να ρωτήσω για αν μπορεί να μου διευκρινίσει κάτι για τις ε, ψηφιακές πλατφόρμες σε περιφερειακό επίπεδο. Όλος ιδιαίτερο σε σχέση με τις λειτουργίες που θεωρεί ότι θα μπορούσαν να έχουν αυτές οι πλατφόρμες. Είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον για μας που εργαζόμαστε για τη συνοχή και τις περιφέρειες και να σκεφτούμε πώς μπορούν να έχουν μια συμπληρωματική στατικική στο ψηφιακό κλάδο ε, οι περιφέρειες, στηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όλους τους φορείς. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε κύριο Χάουαρτ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι πολύ ενδιαφέρον ακαδημαϊκό πόνημα αυτό που είδαμε και διέτρεξα τις 69 σελίδες κάπως εντάχει. Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα που θα μπορούσαμε να τα σκεφτούμε και να τα μελετήσουμε περαιτέρω, αλλά υπάρχει κάτι που κάπως με ξενίζει σε πρώτη αντίδραση στο έγγραφο αυτό για το πώς ε, θα κατευθύνουμε την υλοποίηση. Έχω πραγματικά πρόβλημα όταν το σκέφτομαι αυτό, διότι στην πράξη τι θα σήμαινε για τις επενδύσεις ε, στις ε, εταιρείες τεχνολογίας. Δεν είμαι 100% πεπισμένος ότι απλά μπορούμε να λάβουμε μια απόφαση που θα λέει αυτό θα το κάνουμε στα πλαίσια της περιφερειακής πολιτικής και θα χρησιμοποιήσουμε στην πολιτική συνοχή ως κινητήρια δύναμη της ε, τεχνολογίας. Ακούγεται πολύ ωραίο, αλλά χρειάζονται κάποια κριτήρια επιτυχίας και αυτό που πραγματικά δεν βλέπω από αυτή τη μελέτη είναι τίποτα φοβερά παραδείγματα. Ίσως να μου διέφυγαν, μπορεί, αλλά δεν βλέπω καλά παραδείγματα του τι επιτυχία είχαν όλα αυτά στην πράξη και τι ε, ενδείξεις έχουμε για το πώς μπορεί να είναι αποτελεσματικά αυτά με την περιφερειακή πολιτική. Διότι εάν θέλουμε αυτά τα επιστημονικά κέντρα, τα κλάστερ και οι πυρήνε αυτοί ε, να λειτουργήσουν, χρειάζονται ερευνητέ, επιστήμονε και πρώτε ύλε επιστημονικού χαρακτήρα που να συγκεντρωθούν για να έχουν επιτυχία και σε ένα περιβάλλον αγοράς, αξιοποιώντας αυτά τα βασικά συστατικά που ήδη υπάρχουν. Εάν μιλάμε για πολιτική συνοχή, πού είναι αυτά τα σημεία ε, πού είναι οι πρώτε αυτέ ύλε, πώ θα διοργανωθούν στα επταετή προγράμματα, ε, περιόδου προγραμματισμού. Και για να είναι επιτυχή, χρειάζονται και πραγματικέ επενδύσει σε μικρομεσαίε κάτι σαν αυτό που έχουν στη ΣΥΠΑ. Ε, ένα ενεργότερο κεφάλαιο κινδύνου που μπορεί ο χώρος των επιχειρήσεων να προτείνει ως δευτερογενή μορφή επενδύσεων. Εδώ λοιπόν ε, θα έπρεπε να επικεντρωθούμε στο δεν χρειάζεται να κάνει η ευρωπαϊκή βιομηχανία για να έχει ένα πραγματικό ε, κεφάλαιο κινδύνου για τι επιχειρήσει που μπορεί όντω να στηρίξει τον ιδιωτικό τομέα με επιχειρήσει. Που μπορεί να σύρει όλη αυτή την προσπάθεια, να την οδηγήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκεί θέλουμε να οδηγηθούμε. Και μακροπρόθεσμα πρέπει να καταλάβουμε ότι πολλές από αυτές οι εξελίξεις στην τεχνολογία και τις εταιρείες που ασχολούνται με τις τεχνολογίες ε, κάνουν καινοτόμε μεν ε, λύσεις, προ, προωθούν καινοτόμες λύσεις, αλλά πουλούν προϊόντα όπου παράγουν τεχνολογικές λύσεις ε, και πρωτοπορίες με σκοπό να αγοραστούν τα εργαλεία αυτά που προτείνουν και οι εφαρμογές προτού καν δημιουργηθούν. Αυτό συμβαίνει στη ΣΥΠΑ, ε, εξαγορά των ε, λύσεων προτού καν φτάσουν στην αγορά. Η εταιρεία λοιπόν εξαγοράζεται πριν καν παράγει. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς όλα αυτά μπορούν να συγκεντρωθούν και πού έχουν οδηγηθεί από την αγορά οι όλες οι εταιρείες. Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα επιφυλακτικό για το πώ αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μάλιστα αποτελεσματικά στην πολιτική συνοχή. Ε, συνοχής. Ίσως και να είναι δυνατόν, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί σε σχέση με τα που προτείνει η έκθεση με κριτήρια επιτυχία. Και αν βλέπουμε ε, πράγματα όπω η Ευρώπη μπορεί να τα κάνει αυτά καλύτερα από την Αμερική και την Κίνα, ε, ναι, αλλά πρέπει να ξέρουμε και γιατί και να μπορούμε να απαντήσουμε την ερώτηση αυτή. Δεν βλέπω ε, πού προκύπτει η απάντηση στην έκθεση αυτή. Ευχαριστούμε κύριε Ροπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι το θέμα που μας απασχολεί σήμερα είναι επίγον. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση της μελέτης και συμφωνώ με τους συναδέλφους Και είναι σαφές ότι έχουμε ένα με δύο χρόνια το πολύ για να προετοιμαστούμε για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Κάτι που θα προκαθορίσει το πώς ε, θα λειτουργήσουμε μέχρι τα τέλη της επόμενης περίοδου, τα τέλη του 2028. Σίγουρα μου άρεσαν μερικά σχόλια των συντακτών της μελέτης ότι δηλαδή θα πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τη φιλελεύθερη αρχή κατά την κατανομή των κονδυλίων ή να εφαρμόσουμε αυστηρότερους μηχανισμούς ελέγχου για τον προσδιορισμό των δικαιούχων των κονδυλίων αυτών. Αν κατάλαβα καλά, εσείς είστε υπέρ ε, αυστηρότερων μηχανισμών ελέγχου. Όταν μιλούμε τώρα για την ψηφιοποίηση και την ευφυή ειδίκευση, από πού θα ξεκινήσουμε, ποια θα είναι η αφετηρία μας. Κάποια περίπλοκα προγράμματα ή η εξασφάλιση προηγουμένως της ευρυδονικότητας. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σωστό. Αν εξασφαλίσουμε ευρυζωνικό ίντερνετ και πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε και με νέες πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε την, τον υπερβολικό πειραματισμό. Και να δούμε τα, τα προγράμματα ψηφιοποίησης, όπως ε, το πρόγραμμα για την ηλεκτρονική υγεία, e-health. Κάθε κράτος έχει το δικό του πρόγραμμα με διαφορές μεταξύ των εθνικών προγραμμάτων. Και δεν είναι σαφές αν ο κόσμος ε, έμεινε ικανοποιημένο από τέτοια προγράμματα. Μήπως ε, θα πρέπει πρώτα να καταρτήσουμε κάποιες προτεραιότητες, να δούμε ποιες πρωτοβουλίες θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε κατά προτεραιότητα και να μην ενδιαφερόμαστε μόνο για την απορρόφηση των κονδυλίων και να κάνουμε κάτι τον υστέρων να διαπιστώνουμε ότι κάποια άλλη χώρα το έκανε με καλύτερο τρόπο. Ίσως θα πρέπει να είμαστε πιο επιλεκτικοί στον καθορισμό των προτεραιοτήτων μας και να αποφύγουμε, επαναλαμβάνω, το, την επιπόλαιη ενασχόληση με τον πειραματισμό. Πρώτα να αξιοποιούμε τα κεκτημένα άλλων περιφερειών. Επίσης, μιλήσατε για την ανάγκη να εμπλέξουμε πιο ενεργά τις περιφέρειες. Και εγώ έχω εμπειρία περιφερειακή και πιστεύω ότι ένας τρόπος για να αναμίξουμε πιο ενεργά τις περιφέρειες είναι να μεριμνήσουμε ή τα κονδύλια που δίνονται στις περιφέρειες και στις πόλεις να προέρχονται από τα φορολογικά έσοδα. Κυρίως. Και όταν μιλούμε για εκ των προτέρων αιρεσιμότητα, να εξακριβώσουμε κατά πόσο οι Δήμοι μπόρεσαν να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία μέσω των καλών προγραμμάτων που δρομολόγησαν. Θα πρέπει να γνωρίζουν ε, ότι θα καρποθούν ένα τμήμα της προστιθέμενης αξίας. Και αυτή θα είναι η ανταμοιβή του. Φυσικά οι περιφέρειες είναι διαφορετικέ και δεν θα πρέπει να έχουν όλε τι ίδιε δραστηριότητε και τα ίδια προγράμματα. Πάντω σημαντικό θα ήταν στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού να καταρτήσουμε με σαφήνεια τις προτεραιότητες και να έχουμε ειδίκευση με κονδύλια που θα χρηματοδοτούν σαφώς προκαθορισμένες προτεραιότητες για να μην έχουμε κατανομή κονδυλίων που δεν θα μας εξασφαλίζει επιθυμητά αποτελέσματα. Και δεν είναι ένα καλό παράδειγμα αποκεντρωμένης διαχείρισης των κονδύλιων, ένα αποκεντρωμένο κράτος. και εκτεταμένης εφαρμογής της επικουρικότητας. Και όταν μιλούμε για την επόμενη περίοδο της πολιτικής συνοχής, θα πρέπει να έχουμε υπόψη και αυτές τις αρχές της αποκέντρωσης και της επικουρικότητας. Αυτές οι δύο αρχές είναι πολύ σημαντικές και θα πρέπει να εφαρμοστούν και στο μέλλον. Έτσι θα θερύνουμε και τις τοπικές και περιφερειακές ε, κοινότητες να εμπλακούν πιο ενεργά. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συντάξει τη εξαιρετική έκθεση και θα ήθελα να σχολιάσω για δύο, δύο πράγματα τα οποία διευκρινίζονται στην έκθεση. Η κατάσταση αφορά τις περιφερειακές και τοπικές αρχές θα πρέπει να βρεθούν ε, οι τρόποι ε, συνεργασίας μεταξύ περιφερειακών και τοπικών αρχών. Στο παρελθόν, πολλές ε, χώρες είχαν λυπή συνεργασία. Και νομίζω ότι θα πρέπει να γνωριστεί καλύτερο ο ρόλος των ε, περιφερειακών αρχών και να συμμετέχουν στο σχεδιασμό των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής. Θα πρέπει να δουν κίνητρα στις χώρες μέλη, μέλη ούτως ώστε να ε, προωθηθεί κάτι τέτοιο. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά τον προσεχή γύρω χρηματοδότησης της ε, περιφερειακής πολιτικής. Το άλλο το οποίο αναφέρατε ε, τι I think, uh, companies would have started... Είναι η θερμοκριτήρια των επιχειρήσεων. Ε, νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις μικρές ε, επιχειρήσεις και θα πρέπει να δούμε πώς εξελίσσονται και κατά πόσο επίσης ε, μπορεί να γίνει συνεχή μια επιτυχία με τα science parks. Ε, νομίζω ότι θα μπορούσαν να διαμορφωθούν καλύτερα εάν υπήρχε άμεση διασύνδεση με τα πανεπιστήμια και τα επιστημονικά κέντρα. Ε, νομίζω ότι αυτό ήταν από τα καλύτερα νομίζω ότι από τα καλύτερα παραδείγματα μπορούμε να έχουμε είναι στην Κίνα αλλά και στην Ευρώπη ε, εφόσον υπάρχει αυτή η σύνδεση των ε, επιστημονικών πάρκων με τα πανεπιστήμια. Μελλοντικά λοιπόν, στο πλαίσιο πολιτικής συνοχής θα πρέπει να μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε αυτές τις διασυνδέσεις μεταξύ των science parks και των ε, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ούτως ώστε να υπάρξουν συνέργειες και να δούμε τι γίνεται μελλοντικά όσον αφορά την χρηματοδότηση της κοινωνικής ε, ανάπτυξης. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχυθούν αυτές οι δύο συνδέσεις, όπως σας είπα. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ε, ευχαριστούμε για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καθηγητά, κύριε Άνεστετ, ε, είστε έτοιμος για να απαντήσετε τις ερωτήσεις, να σχολιάσετε απάντηση «Όχι, <laughs> δεν είμαι έτοιμος». Ε, πρόκειται για ένα ευρύ φάσμα πολύ σύνθετων ε, ζητημάτων τα οποία τέθηκαν και τα οποία είναι, παραμένουν σημαντικά, έχουν τέθηκε στο παρελθόν, ε, παραμένουν σημαντικά και θα παραμείνουν σημαντικά. αυτό δεν είναι πρόσχημα για να μην καλύψω όλα τα θέματα αλλά είναι δύσκολο να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ αυτού που κάνει κανείς όταν έχει αυτή την προσέγγιση της δυναμικής ε, τοποθέτησης ε, και θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσαρμόσιμος, αποτελεσματικός ε, όσον αφορά την ανάπτυξη πολιτικής εφαρμογής. και θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα αναγκαία εργαλεία όσον αφορά τον έλεγχο της χρηματοδότησης. Ε, στο επόμενο σημείο της μέσης της διάταξης, ο Φέρη θα σας πει κάποια πράγματα σχετικά ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά την αξιοποίηση των χρημάτων και το θέμα της αποτελεσματικότητας σύμφωνα με τα όσα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και Περιφερειών. Ε, στο του τελευταίου θα πρέπει να βρούμε ένα ευρύτερο πλαίσιο και ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο για τις περιφέρειες και τις επιχειρήσεις ε, που λειτουργούν στο επίπεδο αυτό. Θα πρέπει να υπάρξουν λίγο περισσότερα ανοίγματα, ώστε η περίφημη ευελιξία για την οποία μιλούμε να είναι πιο προσαρμοστική, να είναι πιο στραμμένη προς το μέλλον, να, είναι πιο... να υπάρχει ετοιμότητα να ληφθούν κάποια ρίσκα. Ε, όσον αφορά τις διαδικασίες ε, καινοτομιών και να υπάρχει και μια συνεργασία με τον δημόσιο τομέα. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν με αυτή η σωστή υπεσορροπία. Αυτό είναι μια πρόκληση για όλους μας, όχι μόνο για τους επιστήμονες αλλά και τους πολιτικούς. Να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε ένα αποτελεσματικό σύστημα όπως τις ΣΥΠΑ και άλλα μέρη του κόσμου όπου δίνεται μεγαλύτερη, ε, μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών ε, στους επιχειρηματίες και χειρισμών χωρίς να υπάρχουν όλοι αυτοί οι καταναγκασμοί στον ιδιωτικό ε, τομέα. το να βρούμε αυτή την ισορροπία, να βρούμε αυτή την, μια, έναν άλλο τρόπο λειτουργίας, αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλιώς το σύστημα θα είναι πολύ άκαμπτο και θα καταλήξουμε σε μια επένδυση πολλών χρημάτων εδώ χωρίς να έχουμε τα αναγκαία ωφελήματα. Και θα ήθελα να θυμίσω επίσης το εξής, τα συστήματα τα οποία συγκρίνονται με τις ε, Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ ο, ενεργός, ο δημόσιος τομέας είναι πολύ ενεργός όσον αφορά την ε, προμήθεια χρημάτων στον ιδιωτικό τομέα για καινοτομίες. Για παράδειγμα, στα πανεπιστήμια από το Πεντάγωνο ή από το Υπουργείο Αμήνης. Η χρηματοδότηση επιτρέπει εδώ να γίνουν πολλά πράγματα υπό τη μορφή της χάραξης μιας βιομηχανικής πολιτικής η οποία παρέχει στην κοινωνία, στα πανεπιστήμια και τον ιδιωτικό τομέα πολλά χρήματα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Και επιπλέον έχουμε έναν ιδιωτικό τομέα εδώ ο οποίος πραγματικά στηρίζεται σε αυτή τη χρηματοδότηση γιατί όταν ε, η κυβέρνηση των είπα ε, δίνει πάρα πολλά χρήματα, ε, χρήματα στο, στη Silicon Valley προκειμένου να γίνουν αυτές οι κοινέ επενδύσεις. Αυτό δεν συμβαίνει στην ε, Ευρώπη με τον ίδιο τρόπο, αλλά μπορούμε να βρούμε άλλους τρόπους πιο διαφανείς, πιο ανοιχτούς κλπ. Η απάντηση λοιπόν είναι, στην κυρία Κλάρη, ότι οι προϋποθέσεις πλαίσιο θα πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρες ε, και θα πρέπει να βρεθούν τα ανοίγματα προς τους επιχειρηματίες στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι θα πρέπει να, ούτως ώστε να συνεργαστούν. Ε, παραδείγματα στις τεχνολογίες των ιατρικών συσκευών. Εδώ βλέπουμε σημαντικά πράγματα να γίνονται στην Ευρώπη. Ε, που υπάρχει ένας συνδυασμός ψηφιακής τεχνολογίας με άλλους τύπους τεχνολογιών και ε, τέτοιου είδους επενδύσεις στον τομέα της υγείας με ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Και εδώ βλέπουμε ότι ο δημόσιο τομέα είναι πολύ γενναιόδωρο, παρέχοντα στα νοσοκομεία, πανεπιστήμια, μέσω τη χρηματοδότηση των περιφερειών και εστιάζοντα σε τέτοιου τύπου συνεργασίε σε συγκεκριμένε περιοχέ, υπάρχουν πολύ πετυχημένα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, όσον αφορά τα ακουστικά, ε, ε, στη δική μου χώρα, συσκευέ αυτές, τα βοηθήματα ακοής. Εδώ ε, η Δανία ε, είναι ηγείται γιατί ακριβώς έγινε μια πετυχημένη σύζευξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέας παρέχοντας τα μέσα για τον ιδιωτικό τομέα και σε συνεργασία με το δημόσιο τομέα προκειμένου να φτιαχτούν, να κατασκευαστούν αυτές οι, αυτές οι συσκευές, αυτά τα βοηθήματα για την ε, ε, ακοή, τα ακουστικά. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα περιθώριο ελιγμών εφόσον βρούμε το σωστό επίπεδο ανοιγμάτων. Αλλά το θέμα αυτό είναι πολύ βέστητο και βέβαια χρειάζεται και μια, ένας επαγγελματικός προβληματισμός, όχι μόνο από τους πολιτικούς αλλά και από τους ε, ε επιχειρηματίες και τους εμπειρογνώμονε. τους ειδικού. Ε, και πιστεύω ότι πολλά πράγματα θα μπορούσαν να συμβούν όσον αφορά την πολιτική συνοχή και τι περιφέρειες προκειμένου να βρεθούν τα πιο ειδικά δυνατά σημεία των περιφερειών. Οι πόλεις μας, μας χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, οι υπηρεσίες των, ε, των πόλεων θα πρέπει να ενισχυθούν, υπάρχουν οι τεχνικές λύσεις, αλλά θα πρέπει να ε, μεταφερθούν στις ε, κοινωνικές ποιες καινοτομίες οι οποίες ε, απαιτούνται να αναπτυχθούν στο επίπεδο των περιφερειών με τους διαθέσιμους πόρους. Μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα και θα μπορούσα να σας απαριθμίσω ένα φα... ευρύτερο φάσμα στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών κλπ. Όλοι οι τομείς αυτοί είναι ανοιχτοί για μεταβολές και βελτιώσεις προκειμένου να υπάρξουν νέες ε, λύσεις ε, ύψης της για τους ε, πολίτες και ενδιαφέρουσες και για τους επιχειρηματίες προκειμένου επίσης να, υπάρξουν, να γίνουν και εξαγωγές και στις άλλες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθούν να βρεθεί στο μείγμα μεταξύ των, της ανάγκης ελέγχου και διαφάνειας να τη χρηματοδότηση και της ανάγκης ύπαρξη ευκαιριών για τους επιχειρηματίες και για τις καινοτομίε στο δημόσιο τομέα προκειμένου να λειτουργήσει αυτό το νέο πλαίσιο. Χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια όσον αφορά την ε, πολιτική συνοχής ε, με αυτό τον ε, ενεργό και τρόπο λειτουργίας με ένα πιο ενεργό τρόπο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ηλεκτροντικά έντυπα από την τωρινή συνεδρίαση έχουν link για την έκθεση και μπορείτε να την τυπώσετε και όλες για να την έχετε και σε τεύχος. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ε, όλη παρουσίαση και συζήτηση και ε, σε άλλη ευκαιρία ευχαριστώ να σας υποδεχτούμε και πάλι στην Επιτροπή μας. Και τώρα να συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη παρουσίαση μελέτης που παρήγγειλε η Υπηρεσία Πολιτικής Β για τον έλεγχο και την απλούστευση των διαδικασιών εντός των διευθυντικών και επενδυτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την έκθεση αυτή την ε, ζήτησε η Επιτροπή Ρέτζη και την παρήγγειλε η Υπηρεσία Πολιτικής για τις Διαδοτικές και Πολιτικές Συνοχής με γενικό στόχο να αξιολογήσει τη σχέση μεταξύ των δύο συνιστοσών των Ευρωπαϊκών Επενδυτικών και Διαδοτικών Ταμείων για τον έλεγχο και τα συστήματα ελέγχου και για την μέτρα απλούστευσης που έχουν σχεδιαστεί για να μειώσουν την, ε, και να περιορίσουν την περιπλοκότητα της υλοποίησης του ΕΣΥ. Την παρουσίαση θα μας κάνει ο ε, αρμόδιος ερευνητής κ. Μάρτιν Φέρι από το Κέντρο Μελετών για τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde του Ηνωμένου Βασιλείου. Να δώσω το λόγο στον κύριο Φέρι. Και μετά οι συνάδελφοι θα μπορέσουν να σας θέσουν ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ η μελέτη μας. Μελετά τη σχέση μεταξύ των δύο συνιστοσών των Ευρωπαϊκών Διευθυντικών Ταμείων και των Επενδυτικών Ταμείων για να δούμε κατά πόσον τα συστήματα ελέγχου και τα μέτρα πλούστευσης έχουν περιορίσει την περιπλοκότητα στην υλοποίηση. Θέλουμε να αναλύσουμε τη σχέση για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και τις επιδόσεις, κάτι που είναι σημαντικό και για τη μεταρρύθμιση του ΕΣΥΦ. Οι πρόσφατε προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΣΥΦ στο νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο σκοπό έχουν να βελτιώσουν την ε, οικονομική του διαχείριση αλλά και το πεδίο και την περιπλοκότητα και το άχθο για τους δικαιούχου, δηλαδή του φορείς που εφαρμόζουν και πρέπει στην ε, δημοσιονομική του διαχείριση να εντάξουν και τα του ΕΣΥΦ. Εδώ λοιπόν αναθεωρήσαμε και επισκοπήσαμε τα ωφέλη και πλεονεκτήματα τις σχέσεις μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων και μετά θα δούμε και τι γίνεται μετά το 2020, ολοκληρώνοντας με κάποια συμπερασμάτα και συστάσεις. Ως προς τη μεθοδολογία και τους ειδικούς στόχους τους αναφέρει η διαφάνεια αυτή, η μεθοδολογία μας συνδύασε μελέτη παραδειγμάτων και συνεντεύξεις από ε, ευρωπαϊκά κράτη, επτά συγκεκριμένε υποθέσει με ε, μείγμα ε, προγραμμάτων ΕΣΥΦ. Μιλήσαμε με αρχές διαχείρισης και αρχές ελέγχου από επτά κράτη-μέλη. Πολύ σύντομα να συνοψίσω τα ωφέλη και το κόστος σε σχέση με τον έλεγχο και τα συστήματα ελέγχου των προγραμμάτων ΕΣΥΦ. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε τον ειδικό ρόλο των ελέγχων ε, για το ΕΣΥΦ για να ενισχύσουν την ε, αποδοτικότητα και την λογοδοσία του συστήματος διαχείρισης του ΕΣΥΦ. Υπό αυτό το μοντέλο η λειτουργία των συστήματων αυτών είναι ευθύνη των αρχών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο σημαντικό μερίδιο του ευρωπαϊκού προλογισμού κατευθύνεται προς τα εδώ, οπότε τα σφάλματα στη χρηστή διαχείριση του ΕΣΥΦ είναι σημαντικό να αποφεύγονται. Και τρίτον, υπάρχουν και οικονομικά ωφέλη, τα οποία είναι προφανή για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και τα οποία επιβάλλουν να εντοπίζουμε ατασταλίες ή ε, κακοδιαχείριση για να έχουμε καλύτερη χρήση των κονδυλίων. Οι διαδικασίες απλούστευσης έχουν βελτιώσει την ανείχνευση και διόρθωση των ε, ε, κακοδιαχειρήσεων για να βελτιωθεί συνολικά η υλοποίηση των προγραμμάτων. Οι εμπειρίες από το 2013 και μετά έως το 2017 ε, βλέπουμε μια σειρά από δικαιούχου. Πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποίησε τι οικονομικέ διαχειρήσει για να προστατεύσει διορθώσει, για να προστατεύσει τον ευρωπαϊκό προπολογισμό σε σχέση με το παρελθόν, με μέτρα όπως αναστολή, ε, διακοπή πληρωμών, αναθεωρήσεις, πράγματα που ε, εφαρμόστηκαν νωρίτερα ε, και επιτρέπουν την εγκαιρότερη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης. Όλοι μας έχουμε βελτιώσει τα προγράμματα αυτά με μεγαλύτερο και καλύτερο αποτέλεσμα στο ποσοστό σφάλματος. Επίσης, έχουμε περισσότερη και καλύτερη αντιμετώπιση των δυσκολιών. Βλέπουμε ότι έχουμε προχωρήσει στην ε, σωστό έλεγχο των κεφαλαίων, στην ε, στο 2016 στον σωστότερο καθορισμό και στην αντιμετώπιση του υψηλού διοικητικού κόστους. Αυτό έχει περιορίσει τον αντίκτυπο ε, στα προγράμματα ΕΣΥΦ. Εδώ ε, μπορεί να έχουμε λοιπόν ε, λιγότερα κίνητρα για ε, επικίνδυνες και πιο δύσκολες περιπτώσεις και για ορισμένους δικαιούχους. Εδώ λοιπόν πρέπει η ποιότητα να μας απασχολήσει περισσότερο και να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την κακοδιαχείριση. Στην Στη διαφάνεια αυτή θέλω να περάσω σε περισσότερες ε, λεπτομέρειες για το περίπλοκο σύστημα με τις πολλές διαδικασίες και τους πολλούς ε, φορείς που εμπλέκονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικό. Η διαφάνεια αυτή αναφέρει τις βασικές αρμοδιότητες ελέγχου των αρχών στα κράτη-μέλη, τις αρχές διαχείρισης, ε, τις αρχές που εμπλέκονται στο όλο σύστημα ελέγχου για κάθε πληρωμή ΕΣΥΦ, τους επιτόπιους ελέγχους των δικαιούχων ε, και τις αιτήσει αναθεωρήσεις με τις εκθέσεις και τα μέτρα καταπολέμησης της απάτης. Οι αρχές οφείλουν να υποβάλουν έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να, καταρτήσουν, να διεξάγουν έλεγχο για τη συγκεκριμένη πληρωμή, να οργανώσουν τους ορκωτούς ελέγχους και να συντάξουν επίσης και άλλη σχετική έκθεση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Διευθυντήριο του ΕΣΥΦ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει την κατάρτιση εκθέσεων. Επίσης υπάρχει ο έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο που κάνει τον έλεγχο για τα κονδύλια που το Κοινοβούλιο και το πλαίσιο. Και εδώ γίνονται οι ανάλογες εκθέσεις ε, ορκωτού ελέγχου για όλες τις ε, διαδικασίες. Προσπαθήσαμε να ε, εντοπίσουμε πού είναι πιο περίπλοκες οι διαδικασίες. Από διαφάνεια αυτή βλέπετε ότι η δυσκολία του καθορισμού των συστημάτων ελέγχου ήταν η βασικότερη για το διάστημα 2014-2020. Για τις αρχές διαχείρισης ε, το βασικό ήταν τι έλεγχος μπορούσε να γίνει την καθημερινή πληρωμή και πώς μπορούσε να πλουστευτεί όλη η διαδικασία. Επί τόπου ε, εξακριβώσεις είδαμε ότι γενικώ δημιουργούν ένα μικρότερο πρόβλημα. Ενώ τα μέτρα κατά πολέμηση της απάτης ήταν δύσκολο να υλοποιηθούν γιατί σε κάποιες περιπτώσεις οι αρχές διαχείρισης έχουν την εντύπωση ότι δεν έχουν και δυναμική βάση για να κάνουν τέτοιου επιτόπιους ελέγχους. Η ετήσια επιβολή εκθέσεων έχει ωφέλει ως προς την διευκόλυνση ε, για το κλείσιμο κάποιων προγραμμάτων και την ολοκλήρωσή τους, αλλά σε μακροπρόθεσμη ε, προοπτική ε, δυσκολεύουν τα πράγματα. Για τις αρχές ελέγχου υπήρχαν δυσκολίες για τη διοργάνωση και των ίδιων αυτών των αρχών ελέγχου, ως προς την, τον καθορισμό μέσω της γνωμοδότησής τους, τη στρατηγική του ελέγχου και την συνεργασία τους με τις αρχές διαχείρισης ε, στο σωστό χρονικό πλαίσιο. Επίσης, ο ετήσιος έλεγχος απαιτεί ένα περίπλοκο σύστημα με την δειγματοληψία για συγκεκριμένε ε, πληρωμές και διαδικασίες, κάτι που καθησυχάζει με τις αρχές, αλλά σε επίπεδο χώρας μπορεί να παρουσιάζει ιδιαίτερη περιπλοκότητα. Και πάλι, η αιτήσεις εκθέσεις ελέγχου φάνηκε να περιορίζουν την περιπλοκότητα και γι' αυτό σε αιτήσια βάση να διοργανώνονται πιο εύκολα. Εδώ βλέπουμε κάποιες περιπτώσεις που έχουν ιδιαίτερη περιπλοκότητα λόγω συγκεκριμένων ε, χαρακτηριστικών τους, όπως ε, οικονομικά προγράμματα ή προγράμματα με ειδικά στοιχεία κάποια κράτη-μέλη έχουν αποκεντρώσει τις αρχές ελέγχου και αυτό έχει διευκολύνει το όλο σύστημα ελέγχου. Κάποιες χώρες έχουν περισσότερη θεσμική σταθερότητα και αυτό διευκολύνει για να αντιμετωπιστεί η περιπλοκότητα όταν οι θεσμοί είναι σταθερότεροι σε βάθος χρόνου. Επίσης, όπως τη διαχείριση, ε, η διαχείριση μπορεί να έχει ε, εκχωρηθεί εξωτερικώς ή τουλάχιστον μέρος των αρμοδιοτήτων διαχείρισης και αυτό να έχει διευκολύνει τα πράγματα. Επίσης, σχέση, ε, σημασία έχουν και οι σχέσεις μεταξύ εγχώριας και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Κατά πόσον η εθνική νομοθεσία δηλαδή επιτρέπει να ικανοποιηθούν οι ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Έτσι περιορίζεται η περιπλοκότητα. Και βεβαίως είναι και το ευρωπαϊκό στοιχείο που μπορεί να επιβαρύνει την περιπλοκότητα. Δηλαδή να υπάρχει το σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο με σωστή καθοδήγηση για τις πιο προβληματικές περιπτώσεις ε, με τις δημόσιες προμήθειες συγκεκριμένα και τους κανονισμούς για τις κρατικές βοήθειες. Ένα φάσμα μέτρων έχουν εισαχθεί το 2013 για να αντιμετωπίσουν μερικά αυτά τα προβλήματα και μερικά άρχισαν ε, να εφαρμόζονται από την ε, αρχή του πίστης περίοδου αυτού. όπως οι γνωτήσεις για τον ορισμό χωρίς επιπλέον ελέγχους από το κάτω μέλος και χωρίς επιπλέον κόστος με καταποκοπή ποσά και με ε, συγκεκριμένο κόστος. Επίσης η αναλογικότητα ε, χρησιμοποιήθηκε για τον ε, υπολογισμό του κινδύνου κάποιες φορές για το κόστος και για μερικά προγράμματα που ελέγχθηκαν επί τόπου. Κάποια απλούστευση έγινε και στα δημοσιονομικά εργαλεία για τα προγράμματα συνεργασίας με τις επιλογές απλουστευμένου κόστους. Σε ό,τι αφορά τις εμπειρίες μας από αυτές τις πρωτοβουλίες για την περίοδο 2014-2020, Κάναμε έρευνα βασισμένη στι συγκεκριμένε περιπτώσει και είδαμε ότι οι πρωτοβουλίε αυτέ είχαν κάποιο καλό αποτέλεσμα συνολικά, αλλά χρειάζεται κάποια περαιτέρω βελτίωσή του. Με καταξωσοδότηση πράξη, εφορμαστικέ πράξει, ε, με καθοδήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα κράτη-μέλη Έχουμε αρνητικά αποτελέσματα των ελέγχων. Οι αρχές διαχείρισης έχουν πολύ δειλή προσέγγιση με ήπια χρήση των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καλύψουν όλες τις ανάγκες τους και με μελλοντικέ διαδικασίες ελέγχου. Οι ρυθμίσεις για τα δημοσιονομικά εργαλεία, όλες αυτές είναι καλοδεχούμενες, αρκεί ειδικέ ρυθμίσεις να εισάγονται με τρόπο προσεκτικό οι επιλογέ απλουστευμένου κόστου επίση είναι καλέ για τι αρχέ και του δικαιούχου, όμω σε πολλέ περιπτώσει χρειάζεται το σωστό χρονικό πλαίσιο και δυνατότητε για να εφαρμοστούν. Νομίζω ότι συνολικά Πολλέ από αυτές τις πρωτοβουλίε, όπως το ενιαίο μοντέλο ελέγχου, ο εθνικό καθορισμό, οι απλουστευμένε επιλογέ κόστου, είναι χρήσιμες, όμως πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως με βάση την εμπιστοσύνη και την χρήση δυνατοτήτων, χωρίς να υπάρχει μεγάλος φόβος για τα μελλοντικά σφάλματα που μπορεί να γίνουν. Επίσης, σημαντικό είναι να σημειώσουμε στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο ότι υπάρχουν και άλλες μεταρρυθμίσεις που προβλέφθηκαν από το 2014 έως 2020 για την αντιμετώπιση της περιπλοκότητας ε, των αρχών διαχείρισης. Ένα παράδειγμα είναι οι κανονισμοί που έχουν ε, να κάνουν με τα στοιχεία του πλαισίου ε, επιδόσεων ή την εξάντερεσιμότητα ή τις εδαφικές επενδύσεις. Ταυτόχρονα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι προσπάθειες απλούστευσης συνεχίζονται. Χαρακτηριστικά παραδείγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η ομάδα υψηλού επίπεδου για την απλούστευση, η ατζέντα για την καλύτερη νομοθεσία και οι προτάσεις όμνιμπους. Σε εθνικό επίπεδο είδαμε ενθαρρυντικά παραδείγματα από τα κράτη-μέλη που αναθεωρούν την εγχώρια νομοθεσία τους για να ευθυγραμμιστούν με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και ορισμένα μείωσαν και τους φόρες προγραμματισμού που ασχολούνται με την υλοποίηση για να βελτιώσουν την πιστοποίηση. Κάποιοι ενισχύουν την επιχειρηματικότητα με στοχευμένη στήριξη προς τους δικαιούχους για να υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης των ε, στοιχείων αυτών. Για το τι θα γίνει μετά το 2020, νομίζω υπάρχουν κάποια βασικά στοιχεία που πρέπει να δούμε. Πρώτα απ' όλα, χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία. Τα διάφορα μοντέλα ελέγχου λειτουργούν σε διαφορετικά πλαίσια ανάλογα με το μέγεθο τη χρηματοδότηση, τι δυνατότητε που υπάρχουν, το κεφάλαιο και δεν έχει χρησιμοποιηθεί, εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο ενίου ελέγχου ή όχι και αν μπορεί να επεκταθεί. Επίση, η οικοδόμηση εμπιστοσύνη και δυνατοτήτων. Τι κριτήρια λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιήσει κανεί για να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στι διαδικασίε ελέγχου. Είναι σημαντικό το ερώτημα και είναι θέμα μια ξεχωριστή ολόκληρη συζήτηση. Η δεύτερη γενική ερώτηση έχει να κάνει με την εναρμόνιση στην ε, χρηματοδότηση, αλλά είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί στην πράξη. Επίσης, σημαντικό είναι να διαφοροποιήσουμε μεταξύ της κατάστασης και της χρήσης των ε, αυστηρών κανόνων του ήπιου ε, μοντέλου και των βελτιστών πρακτικών και ούτω καθεξής. ως προς τα συγκεκριμένα ζητήματα το θέμα είναι ο ρόλος και η εξισορρόπηση μεταξύ των ε, ελέγχων ε, ε, επιδόσεων και αποτελεσμάτων. Ξέρουμε ότι οι επιδόσεις είναι κάτι που έχει διάρκεια και πρέπει να υπολογίζεται διαρκώς, ενώ υπάρχουν και η έλεγχη της οικονομικής συμμόρφωσης, που είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξακριβώνεται και θα πρέπει να το μελετήσουμε περαιτέρω. Επίση, σε πολλά προγράμματα το ε, είδο του ελέγχου που επιλέγεται καθυστερεί την έλεξη των προγραμμάτων. Πρέπει επίση να αναγνωρίσουμε την αναλογικότητα στις ε, λειτουργίες των αρχών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των εθνικών αρχών. Πρέπει να πλουστεύσουμε περαιτέρω με μερικά εργαλεία ιδιαίτερω ε, δημοσιονομικά για την εδαφική συνεργασία και τα σχετικά προγράμματα που είναι παραδείγματα. Πρέπει να πλουστευτούν οι διαδικασίε στατιστική δειγματοληψία από τους αρμόδιους φορείς, η απλούστευση του κόστους να γενικευθεί, αρχίζει να διαδίδεται αυτό περισσότερο, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. και από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που ε, μελετήσαμε, ρωτήσαμε την άποψή τους για το πώς πρέπει να γίνει περαιτέρω απλούστευση. Θεώρησαν λοιπόν ότι πρέπει να γίνει και στην απόδοση κονδυλίων με το ενιαίο μοντέλο ελέγχου, με τον έλεγχο των επιδόσεων, αλλά και τον έλεγχο συμμόρφωσης που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτό το είπαν όλοι καθώς και η υποστήριξη της ε, νομιμότητας της νομοτυπίας και του σωστού, ε, της σωστής ε, δαπάνης. Εδώ η στατιστική, η στατιστική δειγματοληψία εγγυάται την ε, ε, επιτυχία του ελέγχου. Υπάρχουν όμως διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικές μεθοδολογίες. Τέλος η ευελιξία αναφέρθηκε και πρέπει να επιδιωχθεί όπου είναι δυνατό και να ληφθούν υπόψη διαφορετικά είδη διαδικασιών σε διαφορετικούς πολιτικούς τομείς. Αυτό έχει να κάνει με την σαφήνεια και το διαχωρισμό μεταξύ αυστηρών κανόνων αυστηρής νομοθεσίας και ήπιας καθοδήγησης συμβουλευτικής μελετών περιπτώσεων βέλτιστων πρακτικών και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει σώρευση Να ολοκληρώσω επαναλαμβάνοντα τα βασική δυσκολία. Το σύστημα ΕΣΥΦ αρχίζει να είναι όλο και περισσότερο αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση των σφαλμάτων και των κακοφυγηρήσεων. Αυτό όμω μπορεί να ε, διαρκέσει ε, με το ίδιο κόστο και με αντιμετώπιση τη περιπλοκότητα. Είναι σημαντικό να σεβαστούμε κάποιε από τι βασικέ αρχέ που ήδη ανέφερα στην παρουσίασή μου. Εναρμόνιση, σταθερότητα, ευελιξία, συντομία, εμπιστοσύνη, οικοδόμηση δυνατοτήτων. Το χρονοδιάγραμμα είναι επίση σημαντικό και χρειάζεται και ε, βελτίωση στη δικασία των διορισμών, χρήση κάποιου ενίου φορέα ή επιλογής αποστασμένου κόστους, όπου για παράδειγμα ο κανονισμό ΕΣΥΦ δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με καταξιότητα πράξη την αρμοδιότητα να προβλέψει ε, ποσά και καταποκοπήν ποσά για συγκεκριμένε δεξιότητε. Αυτό καθορίζει και την πρόσληψη των επιλογών του απλουστευμένου κόστου. Και καλό θα ήταν η διαδικασία ελέγχου να μην εντοπίσει περαιτέρω κακοδιαχειρήσει και παρατυπίε που θα περιπλέξουν την κατάσταση. Πρέπει να γίνει λοιπόν ένα διαχωρισμό μεταξύ αυστηρών κανόνων, ήπια καθοδήγηση για να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα. Επίσης, ειδικά μέτρα για συγκεκριμένα εργαλεία. Είναι σημαντικό. Χρειάζεται όμως επιότερη καθοδήγηση. για την απλούστευση. Ως προς τις συστάσεις για τους συγκεκριμένους φορείς είναι σημαντικό να συνεχίσει η αναθεώρηση και η βελτίωση των ε, κανονισμών βάσει των αρχών που ανέφερα. Πρωτοβουλίε όπω ε, η ομάδα υψηλού επίπεδου και η πρωτοβουλία, η ατζέντα για την καλύτερη νομοθεσία είναι σημαντικά. Η οικοδόμηση δυνατοτήτων στα κράτη-μέλη είναι επίση σημαντική, όπω η ε, διάδοση των εθελοντικών περιπτώσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, καλώς ε, παρατρύνει τα κράτη-μέλη να ενθαρρύνουν τα κλάστερ να αναλάβουν τις επιλογές αποστευμένου κόστους και να δουν πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία αυτά για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Χρειάζονται πρωτοβουλίες για να υπάρχει καλύτερη συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ανταλλάσσουν αποτελέσματα για τις διαδικασίες και τις ε, ε, επιδόσεις τους. Επίσης χρειάζονται συντονισμένοι έλεγχοι με τις αρχές των κρατών μελών, κάτι που είναι σημαντικό και έχει και θετικές επιπτώσεις. Όπως πρόσφατη μελέτη επιδόσεων από το για τον Τζάσπερ που έγινε σε συνεργασία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Πολωνικής ε, Αρχής Ελέγχου υπό την αιγύδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό ήταν σημαντικό για να βελτιωθεί η διαδικασία πλούστευσης. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και οι παρουσιάσει του στα κράτη-μέλη επίση μπορούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη, την οικοδόμηση δυνατοτήτων και την ε, ε, εξοπιστία. Και αυτό επιτρέπει να Παραμένει το, δικα... το ελεγκτικό συνέδριο μια πηγή ανεξάρτητη ε, συμβουλευτική. Είναι ζωτικός ρόλος του ελεγκτικού συνεδρίου αυτού και θα τον διατηρήσει. Για τα κράτη-μέλη, Παρομοίω είναι σημαντικό να αναθεωρούν συστηματικά την ε, οικία νομοθεσία τους ε, για να αντιμετωπίζουν την περιπλοκότητα. Υπάρχει παράδειγμα από κάτω μέλος όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοίταξε κατά πόσον ε, οι αρμόδιες αρχές είχαν κάνει σωστό έλεγχο των διαδικασιών δημόσιων προμηθειών, αλλά οι εθνικέ αρχέ δεν θεωρούσαν ότι αρκούσε ο έλεγχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκαναν έλεγχο και για τι αρχέ ε, ανάθεση. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό. Πρέπει να υπάρχει και πρωτοβουλία και συμμετοχή των κρατών μελών. Επίση για τα συστήματα διαχείριση και ελέγχου. Πρέπει να δούμε πού μπορεί να ε, υπάρχει περισσότερη απλούστευση με εξορθολογισμό των φορέων και σωστές διαδικασίες υλοποίησης. Τέλος, για τις αρχές ε, προγραμματισμού πρέπει να υπάρχει πρόσβαση για την ενίσχυση των δικαιούχων και την ενημέρωσή τους για να ξέρουν πώς λειτουργεί το σύστημα ΕΣΥΦ. Και αυτό έχει δείξει ότι υπάρχουν ωφέλη σε συγκεκριμένε υποθέσεις όπου αντιμετωπίζετε το σφάλμα καλύτερα βάσει τη ερευνά μα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Thank you, thank you. Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Φέρη για την παρουσίασή σας. Και τώρα ο λόγος στα μέλη της Επιτροπής Ρέγγι. Κύριε Κρέλ πρώτα. Ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ε, πιστεύω ότι εδώ συζητήθηκαν πολλά θέματα που έχουν απασχολήσει και εμάς στην Επιτροπή. Έχω ένα ερώτημα για τη διαδικασία Omnibus που έχει υπάρξει και έχει γίνει σχετική διαπραγμάτευση για την, όσον αφορά την πολιτική συνοχής και το αργότερο τον Ιούνιο και θα, θα ισχύσει μετά την ψήφιση στην Ολομέλεια είναι ο προτινόμενος τρόπος εδώ, αυτός τον οποίο εσείς θα υποστηρίζατε. Θα προτιμούσα μία απάντηση όσον αφορά τα αποτελέσματα της διαδικασίας Omnibus από το να, να τρέχουμε στο παρελθόν και να βλέπουμε τι ισχύει τώρα. Θα πρέπει να στρέψουμε τα μάτια στο μέλλον και αν προτείνει η Επιτροπή η αλλαγή του κανονισμού θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο η πορεία την οποία ακολουθούμε εμείς είναι η σωστή ή τελικά υπάρχουν κάποιες ελλείψεις ή πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση. Ευχαριστώ κυρία Μάλετιτς. Σας ευχαριστώ. Όπως είπε και η κυρία Κρέλ, έχουμε επανειλημμένως εξετάσει αυτή τη δυνατότητα για την απλούστευση. Και κάθε φορά που επιχειρούμε απλούστευση φαίνεται ότι καταλήγουμε σε περαιτέρω περίπλοκη του συστήματος. Πάντως θα πρέπει τουλάχιστον στην επό, στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές όντως να εκπονήσουμε ένα σύστημα που θα είναι πιο ελαστικό, πιο εναρμονισμένο, πιο απλό, ώστε στο νέο κανονισμό να συμπεριλάβουμε και αυτά τα στοιχεία. Αναφερθήκατε στις απλουστευμένες επιλογές κόστους, SEO. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τη δημιουργία ικανοτήτων, γιατί χωρίς τέτοια ικανότητες ε, δεν θα τα καταφέρουν οι εθνικές αρχές. Και μάλιστα οι ευρωπαϊκές ελεκτικές αρχές ε, ε, διαπίστωσαν χαμηλό επίπεδο ατασταλιών, σχεδόν μηδενικό επίπεδο ποστό ατασταλιών, χάρη στις απλουστευμένες επιλογές κόστους γι' αυτό φαίνεται πόσο σημαντικές είναι. Επίσης, από τις εκθέσεις του ελεκτικού συνεδρίου διαπιστώνουμε ότι πάνω από 60% όλων των ατασταλιών αφορούν τη διαδικασία κρατικών προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων. Αυτό είναι ένα χειρότερο μήνυμα προς όλους μας. Θα πρέπει σίγουρα να ενισχύσουμε την εμπειρογνωμοσύνη, την παροχή συμβουλών σε επίπεδο κρατών μελών, ώστε να στηρίξουμε τους τελικούς δικαιούχους και τους εφαρμοστικούς φορείς, να ε, εφαρμόσουν καλύτερα τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, ιδιαίτερα σε εκτεταμένα σχέδια, σε μεγαλεπίβολα σχέδια, γιατί φοβάμαι ότι με το σύστημα αυτό είναι δύσκολη πρόσβαση στον τελικό δικαιούχο και στο, στον εφαρμοστικό φορέα χωρίς ε, ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων. Γιατί θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτά τα υψηλά τα τα στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων και ελπίζω με το νέο σύστημα να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα που είναι και το πιο οξύ. Επίσης, κανένας για τις ε, ε, κρατικές ενισχύσεις ε, και τα θέματα των δημόσιων συμβάσεων είναι οι μεγαλύτερες αδυναμίες στα πιο τροτά σημεία του συστήματος και τα σημεία στα οποία εντοπίζουμε τις περισσότερες ατασταλίες και σφάλματα. Και τέλος, αναφερθήκατε στο πολύ σημαντικό θέμα της εμπιστοσύνης. Mm. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θα πρέπει να έχουμε αμοιβαία εμπιστοσύνη, θα πρέπει να μπορούμε να στηριχτούμε ένα τον άλλον. Και, θα... και δεν είναι πάντα καλό ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, ελέγχουμε τα εθνικά συστήματα ελέγχου και τα εθνικά, οι εθνικές αρχές ε, ελέγχουν τους ε, μεμονωμένους δικαιούχους. Αλλά και οι ιδιωτικοί φορείς θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες δημοσίων συμβάσεων. Γιατί παρόλο που το ποστό συγχρηματοδότηση από τα ταμεία ΕΔΕΤ είναι γύρω στο 30% δεδομένου του επιλέξιμου κόστος και εξαιτία του 30% θα πρέπει οι ιδιωτικοί φορείς να ενημερώνονται για τους κανόνες δημοσίων προμηθειών, δημοσίων συμβάσεων. Και μερικέ φορές είναι να προσπαθούμε να τους προστατεύσουμε από τους ε, αυτούς τους, γιατί στόχος τους είναι να πιάσουν τόπο τα χρήματά τους ε, και χρηματοδοτούν το σχέδιο σε επίπεδο 70%. Οπότε θα πρέπει κάπως να ε, κάνουμε πιο ελαστικούς τους κανόνες και να ενισχύσουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Σας ευχαριστώ κύριε Μάλετιτς. Δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις από την Ομίγυρη, οπότε κύριε Φέρη ξανά έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την πρώτη ερώτηση για την απάντησή μας στις προτάσεις για τον κανονισμό Omnibus. Γενικώ είμαστε υπέρ των προτάσεων του κανονισμού Omnibus. Θέλουμε αξιολόγηση ε, ε, του ενίου ελέγχου, την ε, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Στηρίζουμε τις απλουστευμένες επιλογές κόστους. Θεωρούμε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες είναι αξιόλογες και θα πρέπει να παραταθούν και στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Βέβαια, με ασφαλιστικές δικλείδες και οι ασφαλιστικές δικλείδες είναι η εμπιστοσύνη, η δημιουργία ικανοτήτων, σε μία από τις περιπτώσεις, ε, ή μάλλον σε πολλές περιπτώσεις που εξετάσαμε, είδαμε παρόμοιες διαδικασίες όπου μία, ένα συγκεκριμένο ζήτημα από μία συγκεκριμένη διαχειριστική αρχή του κράτους μέλους υπευλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρότεινε κάποιες κατευθυντήρες γραμμές που υιοθέτησαν και άλλες ε, αρχές διαχειριστικές σε άλλες χώρες μέλη που τις εφάρμοσαν ε, ως ε, κανονισμό. Ενώ ο στόχο ήταν ε, συγκεκριμένες οδηγίες προς την διαχειριστική αρχή που υπέβαλε το σχετικό ζήτημα. Θα πρέπει λοιπόν σίγουρα να εξορθολογήσουμε και να πλουστεύσουμε τα συστήματα, αλλά προσοχή. Θα πρέπει να υπάρχει κανονιστική σαφήνεια, ανάργεια και κάποιος βαθμός εμπιστοσύνης και δημιουργίας ικανοτήτων στα κράτη-μέλη, ώστε όλες αυτές οι χρήσιμες πρωτοβουλίες να εφαρμοστούν και σωστά. Και για το δεύτερο σημείο συμφωνώ απόλυτα με την προλαλή σας και σας ευχαριστώ και για τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και την παρουσίαση που μας κάνατε της μελέτης σας και ευχαριστώ και για τις απαντήσεις. Ολοκληρώσαμε την ημερήσια μας διάταξη. Ένα σημείο μας έχει μείνει μόνο, τα διάφορα. Ερωτώ λοιπόν, υπάρχουν διάφορα. Όχι. Οπότε να σας υπενθυμίσω την επόμενη μας συνεδρίαση που θα γίνει στις 20 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, 9 από τις 9 το πρωί. Και ευχαριστώ και τους διερμήνεις. Ευχαριστούμε και εμείς. Και καλό σας απόγευμα εύχομαι. Λύεται η συνεδρίαση.